Ladies and Καλησπέρα σα, ε, κυρίες και κύριοι. Ε, είναι και ο Μπαρτ Στά. Ε, δεν έχει καθίσει. Τέλο πάντων, καλησπέρα. Χαίρομαι που ήρθατε. Είναι πολύ σημαντική η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν κάποιες ανακοινήσεις έχουμε εγκρίνει την, ε, τα πρακτικά της ε, προηγούμενης ε, συνεδρίασης. Στάλησαν με email, δεν υπήρχαν σχόλια. Όλες οι γλώσσες είναι διαθέσιμες, δυστυχώς όμως δεν έχουμε φιλανδικά. Οπότε και μεταδίδεται βεβαίως η συνεδρίασή μας στο διαδικτύο και περνάμε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο έχουμε το σχέδιο απαλλαγής του Γενικού Προϋπολογισμού της Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, είναι τον λόγο αμέσως στην εισηγήτρια την κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και αυτό το οποίο είπατε. Να σας πω λίγο κάποια πράγματα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο, το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση της Αφρικής, Καραϊβικής και του Ειρηνικού της ε, λεγόμενες χώρες ΑΚΕ δηλαδή, όπως επίσης και των υπερπόντιων κτίσεων. Έχουμε λοιπόν μετά την Συμφωνία Κοτονού την ε, πιο μεγάλη συμφωνία που είχαμε από το έτος 2000 ε, ε, και βεβαίως έχουμε και τη Συμφωνία Σύνδεσης από το έτος 2003. Βασικό στόχο Συμφωνίας Κοτονού είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και αυτό σύμφωνα με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της σταδιακής ένταξης των χωρών αυτών στην παγκόσμια οικονομία. Η Συμφωνία του Κοτονού εκπνέει τον Φεβρουάριο του 2020. Το αργότερο τον Αύγουστο φέτος πρέπει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία. Γι' αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει μια απόφαση εξουσιοδότησης ε, εν ώψη των νέων προκλήσεων ε, που αφορούν την διάθεση των μέλων. Εργάζονται λοιπόν όλοι οι νέες έννοιες ε, της βοήθειας και τη νέα διαμόρφωση του πλαισίου της εξωτερικής βοήθειας. Όλα αυτά θα επιδράσουν στο Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Το Ταμείο ακολουθεί τις αρχές της αηφορίας, της συνοχής και της αποτελεσματικότητας αρχές οι οποίες βεβαίως παίζουν μεγάλη σημασία στο πλαίσιο αυτό της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν και κάποιες βασικές προϋποθέσεις για τον δημοκρατικό έλεγχο και την συνοχή της πολιτικής ε, της ε, Ένωσης, ε, την συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες. Επίσης, σημασία έχει ο συντονισμός για να μειωθεί ο κίνδυνος κατακαιρματισμού, να υπάρχει όσο δυνατόν μεγαλύτερη συνοχή και να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη για τους εταίρους μας. Και βεβαίως σημασία έχει και η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα, καθώς μόνο έτσι μπορεί να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό. Επιτρέψατε μου τώρα να περάσω στην οικονομική διάσταση για την έκθεση απαλλαγής του 2016. 4,2 δισεκατομμύρια από αυτά είναι στο η ΕΕΦ, περίπου τα μισά δηλαδή του ύψους του ταμείου, ενώ 2,2 από αυτά πάνε στο λεγόμενο καταπίστευμα για την Αφρική και 130 εκατομμύρια έχουν δεσμευτεί για το Ταμείο για την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Αυτά τα οποία χρηματοδοτήθηκαν το 2000 από το ΕΕΦ είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε 109 εκατομμύρια ευρώ με 56 πληρωμές. Οι πληρωμές του ΙΕΦ ε, σε έργα με πολλαπλούς πληρωτές είναι γύρω στα 940 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά λοιπόν έχουμε 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία εγκρίθηκαν, 480 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύτηκαν και έχουμε 150 εκατομμύρια ευρώ τα οποία εκταμιεύθηκαν για τα ζητήματα μετανάστευσης. Η έκθεση είναι διαρθρωμένη σε 7 τομείς, ξεκινά με την, διαδικασία, με την διαβεβαίωση αξιοπιστίας και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι αυτή. Οι στόχοι μείωσης ε, κατά 25% των παλαιών ανοιχτών χρηματοδοτήσεων, προχρηματοδοτήσεων ε, κατάφεραμε να επιτευχθούν και είχαμε μία μείωση κατά 36% στο χαρτοφυλάκιο της Γενικής Διεύθυνσης ε, ΔΕΒΚΟ. Έχουμε μια μείωση κατά 15%. Το ελεγκτικό συνέδριο όμως διαπιστώνει πως τα συστήματα ελέγχου και επιτήρησης εξακολουθούν να μην έχουν την αποτελεσματικότητα την οποία θα έπρεπε. Όμως το βασικό είναι ότι το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει πως υπάρχει αξιοπιστία όπως επίσης και η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών και βεβαίως καταφέραμε το ποσοστό του ε, σφάλματος ε, να περιοριστεί στο 3,3% μια ελαφρά πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το δεύτερο αφορά την αποτελεσματικότητα του πλαισίου ελέγχου και εδώ πέρα καταφέραμε να μειώσουμε στο 1,7% το ποσοστό των ε, λοιπόν σφαλμάτων, δηλαδή για πρώτη φορά κάτω από το επίπεδο σημαντικότητας ε, του 2%. Το κόστος του ελέγχου ήταν γύρω στα 208 εκατομμύρια ευρώ το 2016. Το τρίτο θέμα αφορά την διαχείριση του καταπιστεύματος, ε, το οποίο είναι βοήθεια προς τον προϋπολογισμό. υπάρχει ακριβώς εκεί πέρα ο κίνδυνος ε, διαφθοράς ο οποίος πρέπει να περιοριστεί και έχουμε ακριβώς μια εστίαση στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής ε, και φοροδιαφυγής και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού όπως τόνισε η Επιτροπή ε, για τα Panama Papers και βεβαίως ε, να μειωθεί εξάρτηση από την αναπτυξιακή βοήθεια. Κατόπιν έχουμε την απέτηση της ενισχυμένης συνεργασίας με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ε, εδώ πέρα ακριβώς έχουμε μια μεικτή χρηματοδότηση η οποία ελέγχεται ως προς την ε, προσθετικότητά της και ακριβώς έτσι θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος μέχρι το 2030. Το έκτο αφορά την ευθυγράμμιση με τις παγκόσμιες, τις συνολικές αναπτυξιακές προτεραιότητες. Το έχω ήδη αναφέρει και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος ε, στα έργα τα οποία θα είναι φιλικά προς το κλίμα. Το τελευταίο, μια νέα εταιρική σχέση με τις ε, χώρες ΑΚΕ στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030 και μια νέα αναπτυξιακή πολιτική. Επίσης, ε, κατόπιν απέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να περιληφθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στον γενικό προϋπολογισμό. Ε, σε όλα αυτά, λοιπόν, θα πρότεινα να δοθεί η απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για το έτος 2016. Έχουμε ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Οι τροπολογίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 1η Μαρτίου, στην Επιτροπή να ψηφιστούν 19 Μαρτίου και μετά τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία και τους δικούς μας βοηθούς για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν στην ε, σύνταξη αυτής της έκθεσης και ελπίζω πραγματικά να προχωρήσουμε έτσι και στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο τώρα στους και συγητές. Τόμας Δεχόφσκι για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Uh, uh, thank you very much for all... Σας ευχαριστώ για όλη αυτή τη δουλειά την οποία έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με μια έκθεση ENF, από το ENF. Κάποια λίγα προβλήματα παραμένουν με ελάχιστες διατυπώσεις που θα ήθελα να αλλάξουν, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχουμε πρόβλημα με τη δουλειά σας, διότι την ε, φέρατε σε πέρας με εξαιρετικό τρόπο. Την κάνατε πολύ καλά. Θα ήθελα ωστόσο να τονίσω δύο-τρία ζητήματα. Πρώτον, την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια για την, ανάγκη αποφυγής συνεργασίας με τους φορολογικούς παραδείσους, την ανάγκη για μεγαλύτερη λογοδοσία και αξιοπιστία και διαφάνεια για τις δαπάνες, για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια και δεν έχετε πει τίποτα γι' αυτό και τονίζω την ανάγκη να εμπλέξουμε το microfinancing ε, να έχουμε επενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα και να εντοπίσουμε το, να εστιάσουμε στις τοπικές πηγές χρηματοδότησης. Δηλαδή χρηματοδότηση και πίστοση για πολύ μικρές επιχειρήσεις και χρηματοδότηση και πίστοση πολύ μικρής κλίμακας που θα απευθύνεται και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο σε κοινωνικό επίπεδο, θα μετριάσουν ε, το τα προβλήματα που μπορούν να προκαλούνται από τις ε, μεταναστευτικές ροές θα τονώσουν την οικονομία και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη. Η σύνταξη της έκθεσης είναι εξαιρετική και θέλω να σας συγχαρώ για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, στρέφομαι προς το κοινό, υπάρχουν άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής μας που θα, θα ήθελα να πάρουν το λόγο. Εάν όχι, 1η Μαρτίου είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και θα, εγκριθεί, θα υιοθετηθεί η έκθεση στις 19 Μαρτίου στην Επιτροπή μας. Δεν θέλει κάποιο μέλος να ε, θέσει κάποια ερώτηση. Όχι. Μπάρμπαρα, έχεις εσύ το λόγο. Ναι, και εγώ θα ήθελα να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ τον Τόμας. Πράγματι, κάναμε καλή δουλειά με τη δική σας στήριξη. Ήταν ομαδική δουλειά και η γραμματεία συνέβαλε τα μάλα και βεβαίω θα συνεχίσουμε ε, προ αυτή την κατεύθυνση και θα λάβουμε υπόψη μας όλες οι τροπολογίε. Το microfinance, finance, η πολύ μικρή ε, χρηματοδότηση, για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο εξαιρετικά σημαντικό, όπως και η αναλογικότητα και η μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα τα πάρουμε όλα αυτά πολύ σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Προχωρούμε. Έχω ένα τεράστιο κατάλογο ευρωπαϊκών οργανισμών και υπηρεσιών και θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης για τους οργανισμούς αυτούς και τις υπηρεσίες. Ε, ζητώ συγγνώμη για την Ίντρεκτ Καράν που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα, έχουμε το συνεισηγήτη ε, Bart Stas και θα σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε για τους οργανισμούς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Εκπλήσω που δεν υπάρχουν ε, συνάδελφοι παρόντες σήμερα. Δεν ξέρω τι σχέση έχει. Είναι Δευτέρα απόγευμα. Μπορεί. Αλλά νομίζω θα έπρεπε έτσι να το πω με όρους ε, της, ε, του καθολικού δόγματος, ε, έπρεπε να είναι από τις μεγάλες γιορτές σήμερα. Να έχουμε μεγάλη προσέλευση, αλλά τι να πω, ας πούμε ότι είναι Δευτέρα απόγευμα. Λοιπόν, με την ΕΦΣΑ δεν ε, ασχολήθηκα γιατί ε, λόγω του ότι είμαι μέλος σε άλλες επιτροπές ε, έχω ξεκινήσει διαδικασίες κατά της ΕΦΣΑ όσον αφορά την δημοσιότητα των εγγράφων της, οπότε θεωρώ ότι δεν θα ήταν σωστό να αναλάβω και εδώ πέρα την έκθεση. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα ε, κάτι να πω. φαντάζομαι το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι της ΕΦΣΑ. Λοιπόν προσπαθήσαμε να εργαστούμε σοβαρά με την έννοια ότι ξεκίνησα ήδη την δουλειά τον Ιούλιο πέρσι μετά, την, ε, μετά το Στρασβούργο πήρα το αεροπλάνο μέσω Φραγκφούρτης πήγα στην Πολόνια και έφτασα τελικά στην ε, Πάρμα όπου Εκεί πέρα συνεδρίαζαν όλοι οι διευθυντές όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Μια εξαιρετική στιγμή δηλαδή για να τους γνωρίσω όλους ε, για να δούμε και το πώς θα προσεγγίσω το ζήτημα της ε, απαλλαγής ε, όπου είχαμε πραγματικά μια επικοδομητική θα έλεγα διαδικασία και εκεί πέρα είδα θα έλεγα να, χτυπάει η καρδιά των 35 αυτών ε, υπηρεσιών και είδα ποιες ήταν, ποια ήταν και τα προβλήματα τους ε, και ανισχύες τους. Και βεβαίως ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι νομίζω πραγματικά αξίζει να λάβουν τις ευχαριστίες μας για την δουλειά την οποία κάνουν σε πολύ σημαντικά θέματα, κατά το οποίο συχνά υποτιμούμε και πρέπει να το λέμε. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία διαπίστωσα αευθύς αμεσώς ήταν ότι στις επαφές που έχουν με τον έξω κόσμο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι υπηρεσίες αυτές ε, υπάρχει σοβαρή έλλειψη συντονισμού μεταξύ τους. Έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους ε, δίκτυο ε, το οποίο νομίζω παρέχει μια καλή στήριξη όσον αφορά τον συντονισμό αλλά ζητάνε κάποια στήριξη από τα δύο όργανα τα οποία καθορίζουν τον προπολογισμό, δηλαδή το Συμβούλιο Υπουργών και το Κοινοβούλιο. Γιατί ο συντονισμός είναι μια ετήσια συνάντηση των διευθυντών. Όταν μιλάμε λοιπόν για μια υπηρεσία όπως η ΕΦΣΑ ή η υπηρεσία φαρμάκων, δεν είναι εύκολο να διαθέσουν κάποιον από το προσωπικό τους για αυτή την... Είναι εύκολο, με συγχωρείτε, να διαθέσουν κάποιον, αλλά οι μικρότερες υπηρεσίες δυσκολεύονται. Και όπως σας είπα, το διαπίστωσα και εγώ που ήμουν ε, ο ίδιος σε αυτήν την συνάντηση πέρσι τον Ιούλιο, γιατί ακριβώς ε, ε, το θέμα ήταν ποιο θα αναλάβει από πλευρά αυτή η συνάντηση ήταν στην Πάρμα και υποσχεθήκαμε στις υπηρεσίες ότι θα το φροντίσουμε, ότι θα δημιουργηθεί μια επιπλέον θέση, κάποιος ο οποίος θα ασχολείται θα είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης ε, με τον συντονισμό με τις άλλες υπηρεσίες, αλλά αυτό το έπνιξε βεβαίως το Συμβούλιο. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να το πούμε και στην οριζόντια έκθεση ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια θέση συντονιστή των διαφόρων αυτών υπηρεσιών και να καταφέρουμε να πείσουμε και το Συμβούλιο. Λοιπόν, στην προσέγγιση μου για την απαλλαγή ακολούσα την ίδια προσέγγιση που είχα ακολουθήσει και πέρσι όταν ήμουν ε, εισηγητής ε, για άλλες υπηρεσίες και εδώ πέρα βέβαια το πρώτο και σημαντικότερο είναι να δούμε το τι συνέβη στην προηγούμενη απαλλαγή, στην προηγούμενη έκθεση, ποιες ήταν οι παρατηρήσεις που είχαμε κάνει, τι είχαμε ζητήσει από την συγκεκριμένη υπηρεσία και το τι έκανε. Οπότε είδαμε το ερωτηματολόγιο και ακριβώ κάθε έκθεση την οποία υποβάλλω θα δείτε ότι έχει και μία περιγραφή της ε, τρέχουσας ε, κατάστασης. Ακριβώς για να δείξουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά την δουλειά μας, έχουμε μία πολιτική εποπτεία της εξέλιξης ε, των πραγμάτων και παρακολουθούμε το τι γίνεται το δεύτερο το οποίο είχα εισαγάγει και στην έκθεσή μου για άλλες υπηρεσίες είναι κάποια πράγματα τα οποία από δημοσιονομική τεχνική σκοπιά δεν είναι ακριβώς πράγματα τα οποία ίσως αναμέναμε σε μια απαλλαγή, αλλά θεωρώ ότι μια απαλλαγή οπωσδήποτε πρέπει να κινείται και σε πολιτικό επίπεδο. Παραδείγματο χάρη το πώς βλέπουμε μια υπηρεσία από την σκοπιά του performance-based budgeting, όπως ε, λέμε, το πώς ε, δηλαδή ε, χρησιμοποιεί τα κονδύλια. Ένα σημαντικότερο ε, δεύτερο θέμα και πράγματι εδώ πέρα και ο εισηγητής συμφωνεί, το πώς βλέπει η υπηρεσία θέματα διαφάνειας, ε, σύγκρουσης συμφερόντων, τι κάνει με πληροφοριοδότες, αν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός, ε, πώς εφαρμόζεται, αν ε, υπάρχουν προβλήματα ή πράγματα τα οποία δεν είναι ιδανικά και αυτό το είδαμε ξεχωριστά για την κάθε τέτοια υπηρεσία. Το τρίτο δεν θα σας προξενήσει έκπληξη ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ότι κοιτάμε την στελέχωση και το τι γίνεται με μια ισορροπία ανδρών γυναικών. Δυστυχώς ε, ε, βεβαίως ε, υπάρχει μια υπερπροσώπηση ανδρών στις διευθυντικές θέσεις, ενώ γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες αν όχι και καλύτερες ε, ικανότητες και επίσης ε, ε, εντάξει σε μια τέτοια υπηρεσία διαπιστώσαμε ότι ήταν οι άντρες η μειοψηφία ήταν το 1 τρίτο αλλά αυτό ήταν η εξαίρεση γενικά στις, στο σύνολο των υπηρεσιών και προσπαθήσαμε επίσης να δούμε μια πτυχή που θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να βελτιώσουμε την δουλειά των υπηρεσιών αυτών, ε, δηλαδή τι κάνουν για το προσωπικό τους, ε, αν υπάρχουν δραστηριότητες ε, team building, να φροντίσουν να προλαμβάνουν τις ασθένειες, το πώς έχουν συγκεκριμένα δηλαδή τα πράγματα όσον αφορά τις ασθένειες σε κάποιες από αυτές τις ε, υπηρεσίες. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης ε, και αυτό ε, προέκυψε αμέσως στην πρώτη μου επαφή πέρσι τον Ιούλιο στην Πάρμα και μου το έθεσαν οι διευθυντές είναι ο συντελεστής διόρθωσης. Τι είναι αυτό, είναι ένας κανόνας όπου οι ε, μισθοί επανυπολογίζονται με βάση το επίπεδο διαβίωσης ε, της χώρας στην οποία έχει την έδρα του ε, ε, την έδρα της η συγκεκριμένη υπηρεσία. Οπότε προσπαθούν, αλλά είναι ακριβώς δυσκολία να προσελκύσουν προσωπικό όταν η έδρα τους είναι στην Ανατολική Ευρώπη γιατί αυτό σημαίνει έναν μισθό 60% αυτού ο οποίος εργάζεται παραδείγματος χάρη στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν, γιατί σε κάποιες ε, υπηρεσίες ε, υπάρχει πραγματική πιεστική ανάγκη να γίνει κάτι για αυτό το θέμα. Να αναφέρω μια συγκεκριμένη περίπτωση, η Frontex ε, με έδρα τη Βαρσοβία, όπου υπάρχει πραγματική δυσκολία να βρουν κόσμο γιατί αντιλαμβάνεστε λόγω αυτού του Ζητήματο το οποίο είπα. Αυτό είναι λοιπόν ένα πρόβλημα και βεβαίως υπάρχει το θέμα του αντικτύπου του Brexit σε κάποιες τέτοιες υπηρεσίες. Ε, κάποιες έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δύο μεγαλύτερες είναι η Υπηρεσία Φαρμάκων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, αλλά υπάρχουν και άλλες που έχουν και παραρτήματα στον Ηνωμένο Βασίλειο, τον Γαλιλαίο παραδείγματο χάρη, το GNSS και οπωσδήποτε στην όλη αυτή η πολιτική συζήτηση για το πού θα πάει η έδρα όταν φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο, οπωσδήποτε ε, για τις δύο μεγάλες υπηρεσίες, ε, την αρχή τραπεζών και φαρμάκων, ε, ακριβώς ο συντελεστής αυτός ο οποίος σας είπα ότι επηρεάζει τον μισθό παίζει μεγάλο ρόλο από ό,τι φάνηκε στις εσωτερικές έρευνες ε, και ερωτηματολόγια του προσωπικού γιατί από ό,τι φαίνεται 90% του προσωπικού στην ε, περίπτωση της υπηρεσίας φαρμάκων δεν θέλει να ακολουθήσει σε μία μετακόμιση γιατί είναι ο συντελεστής όπως σας είπα ε, είναι ζητήματα κοινωνικά, είναι το ότι ε, οι σύζυγοι, οι σύντροφοι έχουν βρει δουλειά στο Λονδίνο και δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Ε, οπότε όπως σας είπα για αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες θα μεταφερθούν αντιστοίχως στο Παρίσι και το Άμστερνταμ υπάρχουν οι δυσκολίες αλλά βεβαίως το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό οδηγεί σε δυσαρέσκεια για το ότι υπήρχαν και ανατολικές χώρες που ήταν υποψήφιες και ε, είδαν ότι έχασαν την ευκαιρία για να πάρουν αυτές ε, τις δύο Τώρα. Ναι, ξέρω ότι ε, μιλάω αρκετή ώρα. Να πω κάποια πράγματα για κάποιες ε, συγκεκριμένες ε, υπηρεσίες. δεν θα αναφερθώ όμως στην ΕΑΖΟ. Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, αφορά την πολιτική του ασύλου. Έχουμε λοιπόν, είχαμε μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών λέω κάτι σχετικά στο σχέδιο έκθεσής μου στις ε, παραγράφους 5 και 6. Το σημαντικότερο εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει ε, μία έρευνα του Όλαφ ε, η οποία είναι σε εξέλιξη για την ΕΑΖΟ, για την υπηρεσία ασύλου. Κάποιες πηγές λένε ότι είναι πολύ σοβαρή η έρευνα αυτή ο διευθυντής της υπηρεσίας ασύλου, ο κύριος Καλντέρα, λέει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό θέμα, αλλά σε ό,τι μας αφορά, τουλάχιστον εμένα ως εισηγητή, έχω τις επιφυλάξεις μου και θεωρώ ότι και το Κοινοβούλιο, Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, μπορεί να πει ότι δεδομένου του ότι υπάρχει μία ανοιχτή έρευνα της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή. Δηλαδή φανταστείτε να δώσουμε απαλλαγή και να έρθει ο Όλαφ και να πει υπήρχε απάτη. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα του Όλαφ ε, φέτος το καλοκαίρι, οπότε μία αναβολή Τη απαλλαγή για το ΕΑΖΟ σημαίνει ότι θα πάμε στο δεύτερο γύρο τον Σεπτέμβριο και μετά να πάμε στην Ολομέλεια του Εκτεβρίου, αλλά καλό είναι να το κάνουμε τότε για να γνωρίζουμε και πώς έχουν τα πράγματα και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της έρευνας του Όλαφ. Λοιπόν, πρόκειται για δημόσια συνεδρίαση εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι ακούνε και οι άνθρωποι των υπηρεσιών, αλλά και οι δημοσιογράφοι. Ε, είναι λοιπόν ευαίσθητο το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω και το λέω αυτό ρητός ε, στη, στην παράγραφο 27 και σε άλλες εκθέσεις, σε άλλες ε, παραγράφους της μου, η ΕΑΖΟ είναι μια υπηρεσία η οποία κάνει υποδειγματικό έργο. Είχα επαφές με συναδέλφους ε, της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ από τη δικιά μου ομάδα και από όλες τις ομάδες και η ΛΥΜΠΕ ασχολείται συνεχώς ε, με το ΕΑΖΟ και εκεί πέρα εκτιμούν πάρα πολύ το έργο της. Και όπως σας είπα αναφέρω στην παράγραφο 27 τον πολύ ενεργό ρόλο που παίζει η ΕΑΖΟ όσον αφορά την πολιτική του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα και στην Ιταλία, την στήριξη που ε, δίνει σε αυτές τις χώρες η οποία εκτιμάται ε, όλος ιδιαίτερος και τον μηχανισμό μετεγκατάστασης από Ιταλία και Ελλάδα για άτομα τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας ε, και έχει οδηγήσει έτσι σε μια πιο αποτελεσματική αντίδραση σε θέματα ασύλου Οπότε όπως σας είπα ε, εκτιμούν πάρα πολύ το έργο τους και το ότι αναβάλλεται ε, ή θα αναβληθεί η απαλλαγή δεν έχει ουδεμία σχέση με την δουλειά που κάνει ο κόσμος είτε είναι εγκατεστημένος στη Μάλτα, στην Ιταλία, στην Ελλάδα τους οποίους εκτιμούμε πάρα πολύ και οπωσδήποτε αυτό δεν σημαίνει ότι δείχνουμε την ΕΑΖΟ με το δάχτυλο. Σχετίζεται μόνο με το ότι υπάρχει μία έρευνα του Όλαφ εξελίξη και δεν μπορούμε οπωσδήποτε να α, λάβουμε μία θέση η οποία μπορεί αργότερα να διαψευστεί. Τώρα, για τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα του συντελεστή διόρθωσης, όπως είπα τα έχω αναφέρει αυτά και για τη Frontex και για την ΕΑΖΟ, και για τη ΣΕΠΟΛ, για το EDC, την Μπέρεκ και, και την ε, Λίζα. Έχω αφιερώσει για όλα αυτά μία παράγραφο ε, έτσι ώστε και εμείς επισήμως ως Κοινοβούλιο να ζητήσουμε από την Κομισιόν μια επανεξέταση του συστήματος για την ε, τραπεζική αρχή και την υπηρεσία φαρμάκων. Πράγματι, εκεί πέρα ζητάμε να υπάρξει μια σωστή εξέλιξη της ε, μετακόμισης ε, σε Παρίσι και Άμστερνταμ. Έχουμε και όντω μεγάλα προβλήματα με την υπηρεσία φαρμάκων σας τα ανέφερα. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα ότι η ενοικίαση του κτηρίου στο Λονδίνο ε, διαρκεί μέχρι την ε, δεκαετία του 2030 και θα πρέπει ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνει νίκη μέχρι τότε. Ε, ζητάω στον εκτισή μου να βρεθεί μια λύση να φροντίσουμε με κάποιον τρόπο να επιληθεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν βεβαίως ε, να πούμε ότι είναι σωστή αυτή η χρήση του χρήματος ε, των φορολογουμένων. Τώρα, για την ε, εύζα του συναδέλφου Τάραντ βλέπω εδώ πέρα ότι βλέπει με τρόπο επικοδομητικό την απαλλαγή της έφσα όπως ε, και οι άλλοι συγητές ε, Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, ε, να δοθεί περισσότερο βάρος στην σύγκρουση συμφερόντων, στο τι γίνεται με πληροφοριοδότες. Να φέρει κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Υποθέτω λοιπόν πως και οι συνάδελφοι θα κάνουν τις ε, παρατηρήσεις τους, αλλά νομίζω σε γενικές γραμμές ο Ίντρεκ Τάραντ έχει συντάξει μια δίκη, θα έλεγα, έκθεση για την Εύσα και γνωρίζω ότι ταξίδεψε και στην ε, Πάρμα για να συναντήσει προσωπικά τον διευθυντή της υπηρεσίας τροφίμων και ε, από ό,τι μαθαίνω ήταν μια πολύ επικοδομητική η συνάντηση. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα σημεία λοιπόν της δουλειάς που έκανα τους προηγούμενους μήνες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μπάρτ. Ο κύριος Σαουάρμα πρώτα από τους κοιόδης συγητές. Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τον συγητή για το έργο του εξαιρετικό, πολύ επαγγελματικό. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον εισηγητή εν όλο στα περισσότερα από τα σχόλιά του για τις ε, υπηρεσίες. Είναι πολύ λογικά και στηρίζονται από την ε, προφανές στα σχόλια και τις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Επί της ουσίας πρώτα. Υποστηρίζουμε την πρόταση του εισηγητού για απαλλαγή για την ΕΑΖΟ, ελπίζοντας ότι θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα από την έρευνα της ΟΛΑΒ μέχρι το φθινόπωρο. Και τώρα μπορώ να σας κουράσω γιατί έχω εδώ ένα κατάστοιχο των πιο σημαντικών ευρημάτων αλλά θα ξεκινήσω με την επιπλέον θέση για το δίκτυο της υπηρεσίας, την υποστηρίζουμε. Θα έχει κεντρική σημασία για τον αποτελεσματικό συντονισμό της δουλειάς και της επικοινωνιακής ε, δράσης της υπηρεσίας και εν προκειμένου επιτρέψτε μου και δεν αφορά αυτή καθε αυτή την απαλλαγή του 16 να συμπληρώσω ότι δεδομένου ότι πολλοί από εμά είχαμε εκφράσει την επιθυμία η διαδικασία αυτή να επιταχυνθεί και να έχουμε πιο νωρίς στην τη διαδικασία τα, τις προτάσεις. Ίσως μπορούσαμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να είναι και το δίκτυο της υπηρεσίας σε θέση σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ίσως πάνω σε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, να δίνει απαντήσεις πιο νωρίς μέσα στον χρόνο. Επίσης, έμφαση θέλουμε να δώσουμε στο ρόλο του δικτύου της υπηρεσίας, εν όλο, εξέταση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότηση παραδείγματι για τις υπηρεσίες, αλλά και γενικότερα για την προετοιμασία του προσεχούς πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί όντως υπάρχει ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ του δικτύου και της Επιτροπής. Επίσης θα θέλαμε ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση στο ρόλο της υπηρεσίας της συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ώψη του Brexit, των, των ε, συνομιλιών για το Brexit ε, και των προσπαθειών για ε, ελαχιστοποίηση των συνεπειών αυτού του ατυχούς γεγονότος και επίσης μαθαίνουμε ότι υπάρχουν εξελίξεις προς τη συνεργασία της υπηρεσίες, της υπηρεσίας για την ε, προκήρυξη διαγωνισμών σε προμήθειες για υλικό και υπηρεσίες. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά και συντονισμός βέβαια από το δίκτυο. Καλούμε τις υπηρεσίες περαιτέρω να συνεχίσουν να εκτελούν τον προπολογισμό τους με βάση τις ε, επιδόσεις και να αξιολογούν τα αποτελέσματα και το προϊόν για τη μεταφορά κονδυλίων που κάθε φορά έχουμε, τα carry-over. Είναι ένα κοινό πρόβλημα. Πάλι όμως θα θέλαμε μια προσέγγιση ισορροπημένη, όπως άλλωστε στα ο εισηγητής. Υποστηρίζουμε την απέτηση του για, μια, για ένα σαφή σχεδιασμό και λογοδοσία για τις πολιτικές δραστηριότητες και πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν διαφοροποιημένα, διαφοροποιημένες πιστώσεις όπου το προτείνει το ελεγκτικό συνέδριο. Ο χαμηλός αντελεστής ε, διόρθωσης. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι ανησυχούν οι υπηρεσίες και σε ένα βαθμό μπορούμε να συμφωνήσουμε ως προς τα προτινόμενα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι διορθωτικοί συντελεστές μπορούν να υπολογιστούν κατά έναν τρόπο που να αποτελούν κίνητρα πιο σημαντικά και για χώρες υψηλού εισοδήματος. Του τουλεχθέντος βεβαίως θα πρέπει και να επισημάνουμε ότι καθώς οι διορθωτικοί συντελεστές ε, συνδέονται με το χαμηλό κόστος ζωής, αγοραστική δύναμη, ε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτισή τους και τα στοιχεία αυτά, κόστος ζωής δηλαδή, αγοραστική δύναμη δηλαδή κτλ. Επίσης, υποστηρίζουμε τις προτάσεις και ιδέες του εισηγητή για την ε, εξέταση σε οριζόντια ζήτηση και γι' αυτό θα θέλαμε και εμείς ε, οριζόντιους ε, δείκτες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Έτσι ώστε να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία, όπως λέει και ο εισηγητής, ο οποίος ταυτόχρονα για τη διαφάνεια όντως μας λέει ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, σωστά επισημαίνεται αυτό. Επικοινωνία, επικοινωνική πολιτική και ορατότητα της, των υπηρεσιών σε σχέση με την κοινή γνώμη και πάλι εδώ υποστηρίζουμε ε, την ε, θετική αποτίμηση των ε, προόδων και βελτιώσεων που διαπιστώνει και ο εισηγητής και επίσης τελευταίο σημείο συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι το διοικητικό βάρος του ελεκτικού συστήματος επιβαρύνει σοβαρά τις υπηρεσίες και άρα σε μια μελλοντική αναθεώρηση του μεσονομικού κανονισμού ελπίζουμε θα υπάρξει δυνατότητα για πιο σαφείς αρμοδιότητες και ευθύνες. Λυπάμαι, λυπάμαι, αλλά δεν βρίσκω τίποτα πραγματικά αρνητικό να πω για τη δουλειά σας φέτος. Κύριε Στάσμα, μην περιμένετε να λυπηθώ εγώ. Και σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Σαουάρμα. Ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία που μόνο αυροφροσύνες ακούμε απόψε και κομπλιμέντα. Ναι, έπρεπε να πω κάτι ακόμα στην αρχή, λέει ο κύριος Εγώρμα. επιτρέψτε μου και να καταγραφεί. Αυτή η διαδικασία, η αιτήσια επισκόπηση από την Επιτροπή τη δική μας είναι η πιο σημαντική δουλειά που κάνουμε. Το να έχουμε όμως παρουσία 20% τι να σας πω, δηλαδή μπορεί να μην είμαι και εγώ κάθε μέρα στις συνεδριάσεις, αλλά αυτή τη μέρα την τόσο σημαντική θα έπρεπε να είμαστε όλοι παρόντες η Πρόεδρος ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ, όπως άλλωστε είπα και το πρωί και ξεκινώντας, ο κύριος Συναστή Μαλή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου να χαρώ κι εγώ τον κύριο Στάς, τον κύριο Ταράντ, για την ε, λεπτομερή και διεξοδική εξέταση των πεπραγμένων των υπηρεσιών. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ακούσει. Επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση, αποτελέσματα καταγράφονται. Για το τελευταίο θα ήθελα να πω δύο λόγια, με σχόλια και προτάσεις συμπλήρωσης. Πρώτον λοιπόν το πεδίο και η δομή της έκθεσε είναι κατάλογο σχέση με την ε, καταγραφή των υπηρεσιών. Είναι κατάλογο γιατί καταγράφει τα πιο σημαντικά στοιχεία των επιδόσεων. Έχει ειδικά κεφάλαια για τη βασική δημοσιονομική διαχείριση και τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων και των βασικών αρχών ε, της οικονομικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης. Ο ετήσιος σχεδιασμός και η έλεγχη των υπηρεσιών θα μας δώσουν μια σαφή εικόνα για τη λειτουργία του 2016. Επίσης, οι νέες υπηρεσίες 2.364 υπάλληλοι και 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν υψηλή ορατότητα στα κράτη-μέλη και επηρεάζουν σημαντικά την ε, χάραξη πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς οτικής σημασίας για τους Ευρωπαίου πολίτες. Στου τομεί που καταγράφει η έκθεση θα ήθελα να προσθέσω την βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, οικονομικά και νομισματικά θέματα και τις ε, σχέσεις με την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Το 2016 λοιπόν είδαμε, σημαντική, είδαμε μια κάποια αύξηση στον προπολογισμό αλλά και το προσωπικό πολλών από τις υπηρεσίες. Πρέπει να καταγράψουμε και τις, τα νέα καθήκοντα με βάση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον αριθμό των επιδόσεων έχουμε μια γενική, ένα γενικό κανόνα, μια γενική προσέγγιση. Εάν δούμε την αξιολόγηση από το ελεγκτικό συνέδριο των νέων υπηρεσιών σε σχέση με το 2016, έχουμε 41 δομές, εκ των οποίων 32 είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες, 6 εκτελεστικές και 3 λοιπά σώματα, λοιποί οργανισμοί. Προϋπολογισμός και προσωπικό στην ε, ε, ενιαία έκθεση καλύπτει και τα 41 αυτά όργανα ή σώματα και εμείς ε, κυρίως πρέπει να δώσουμε προτάσεις για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Εν προκειμένου θα πρέπει να ενοποιηθεί η μεθοδολογία μας με αυτήν του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σε σχέση με τον ενιαύσιο χαρακτήρα του εις δημοσιονομικής διαχείρισης έχουμε ένα υψηλό επίπεδο μεταφορών κοντιλίων σε σχέση με τον αριθμό και για τις περισσότερες από αυτές τις υπηρεσίες. Λόγω του πολιετούς χαρακτήρα ορισμένων προγραμμάτων αυτό καθίσταται βέβαια αναπόφευκτο. Ωστόσο, αυτέ οι μεταφορέ αναδηλώνουν σε πολλέ περιπτώσει δεν προκύπτουν ω αποτέλεσμα κακή διαχείριση ή ελλειπού εφαρμογή. Αντιθέτω, θα πρέπει να ε, και όσο θα πρέπει το ελεκτικό συνέδριο να τι αξιολογεί κατά αυτόν τον τρόπο, κατά κατάλληλο τρόπο δηλαδή. Επίσης ε, υπάρχουν περιθώρια για ασφάλματα σε ορισμένους τομείς σε σχέση με τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς. Βεβαίω θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ των γνήσια κακών επιδόσεων στο τομέα αυτών ή των παρατυπιών που μπορεί λόγω έκτακτων περιστάσεων να προκύπτουν παραδείγματι λόγω σημαντικού εξωτερικού ή εσωτερικού κινδύνου για την τάξη και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όλο. Και επίσης εν τέλει ε, καλώς ορίζουμε την εγκαθίδρυση ενός νομικού δικτύου για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής ε, με μια έκθεση που θα πρέπει να παρουσιάσει όχι μόνο, όχι απλώς να παρουσιάσετε στο κοινοβούλιο, αλλά μέσα σε χρονικά όρια συγκεκριμένα. Σημαντική θα είναι επίσης ε, για την έκθεση αυτή μια αξιολόγηση ποσοτική της δυνατότητας για αντιμετώπιση και πρόληψη διαφθοράς και παρατυπιών σε σχέση με τις υπηρεσίες αυτές. Μια τελική παρατήρηση εκτός κειμένου που διάβαζε ο μιλητής μέχρι τώρα είναι ότι βεβαίως και εμείς υποστηρίζουμε την ΕΑΖΟ, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τραβήξουμε μια γραμμή για το πότε δηλαδή θα μπορέσουμε να λάβουμε την έκθεση της Όλαφ και όπως ήδη είπε και ο κύριος Σαουάρμα μέχρι το φθινόπωρο. Πρώτη αρχές Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουμε δηλαδή την έκθεση για να μπορέσουμε να προβλέψουμε τη σχετική συζήτηση στο χρονοδιάγραμμά μας Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάπελ, τελευταία και μετά θα δώσω το λόγο στους Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή μας ο οποίος αποδεικνύει την ε, μεγάλη και εις βάθος γνώση του και ε, τις ικανότητες του στο θέμα αυτό. Υποστηρίζω απολύτως την έκθεση, είναι πολύ καλή για την νεά η αναβολή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και θετική και συμφωνώ ότι είναι πολύ απαραίτητο να έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να μπορούμε να αξιολογούμε μέχρι ε, κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες και προκειμένου την ΕΑΖΟ. Για το δίκτυο πολύ σημαντικό θα ήθελα να πω ότι μου φαίνεται το δίκτυο μας βοηθά και στην καθημερινή μας δουλειά να παρακολουθούμε αυτή τη διοργανική συνεργασία, τις ε, σχέσεις συνεργασίας και πιστεύω ότι και για τη μελλοντική μας δουλειά αυτή η συνεργασία με συγκεκριμένα κριτήρια θα πρέπει να προσμετράτε σε σχέση με το δίκτυο ώστε να μπορούμε να υπολογίζουμε τι πραγματικά γίνεται. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, προστασία προσωπικών δεδομένων, προστασία δεδομένων κυβερνοασφάλεια, τρία ε, μάλλον προστασία δικτύων και κυβερνοασφάλεια, Ενίσα, ΕΣΑ, και έτσι εδώ έχουμε να κάνουμε με τρεις διαφορετικές υπηρεσίες. Άρα θα πρέπει να διευκολύνουμε, να, ή, να σπρώξουμε προς την ανάπτυξη του είδους δικτύων. των υπηρεσιών που χρηματοδοτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τη δουλειά των υπηρεσιών αυτών και επίσης για την μεταφορά των κονδυλίων. Πιστεύω ότι και αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με την ε, διοργανική συνεργασία και ίσως καταφέρουμε εδώ να την ε, μετατρέψουμε σε ένα κριτήριο ε, απολογισμού, αξιολόγησης της συνεργασίας αυτής. Το Brexit αναφέρθηκε νωρίτερα, τεράστιο θέμα. Είμαι σκιώδη συγκήτρια για την ΕΜΠΑ, για τις τράπεζες και βέβαια μας έχει απασχολήσει ήδη το θέμα αυτό. Είναι τεράστιο το ζήτημα και των ε, μισθωτηρίων συμβολέων που θα εκπνεύσουν ε, μόλις το 2030. Τι θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, πώ θα τα χειριστούμε και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι κάτι το οποίο και για το μέλλον, ε, για μελλοντικέ δεσμεύσει σχέση με ε, μισοτήρια συμβόλαια ή, άλλες, ε, ή άλλα αντίστοιχη, άλλες αντίστοιχες δεσμεύσεις θα πρέπει να προβλέψουμε. Προβλέποντας ενδεχομένω για το μέλλον περισσότερη ευελιξία από ό,τι τουλάχιστον είχαμε σε σχέση με την ΕΜΠΑ. Νομίζω ότι μπορούμε να διδαχθούμε από αυτήν την περίπτωση του Brexit και για το μέλλον, για τον τρόπο με τον οποίο θα διαπραγματευόμαστε τα συμβολία μας στο μέλλον. Ευχαριστώ, κύριο Στεχόφσκι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η έγκριση για τη δημοσιονομική διαχείριση των οργανισμών και των υπηρεσιών είναι σχολείο πραγματικό. Είναι σαν να κάνουμε μεταπτυχιακό κάθε χρόνο. Ε, θέλει πολλή δουλειά και πάρα πολλή έρευνα και ανάλυση. Και συμφωνώ με τον κύριο Σαρβάμα θα πρέπει η παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής μας να θεωρείται εκ των ουκάνευ. Θα έπρεπε όλοι να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση, είναι εξαιρετικά σημαντική. Και εγώ, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ και τέσσερα χρόνια έρχομαι Παρακολουθώ, είμαι σκιώδης εισηγητής για αυτό το ζήτημα των οργανισμών, των υπηρεσιών. Ορισμένα θέματα αναφέρθηκαν. Αυτό οφείλω να το παραδεχθώ και να το ομολογήσω. Κάποια άλλα όμως όχι. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πολύ περισσότερη κριτική. Εάν οι σκιώδη εισηγητές, εμείς δηλαδή, δεν είμαστε αρκετά επικριτικοί και δεν εφιστήσουμε την προσοχή σε τίποτα και τελικά πούμε ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί δουλεύουν και λειτουργούν φανταστικά, ε τότε δεν θα έχουμε συμβάλει καθόλου. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία της απαλλαγής, της έγκρισης των λογαριασμών χρησιμεύει σε πάρα πολλά πράγματα και κυρίως χρησιμεύει στο να τεθούν τα ζητήματα στις σωστές τους διαστάσεις. Όταν ξεκίνησα τη θητεία μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είδα ότι η πλειονότητα των υπηρεσιών και οργανισμών που εδρεύουν π.χ. στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία είναι πολύ λίγες. Για παράδειγμα, να το πω αλλιώ. Οι περισσότερες υπηρεσίες εδρεύουν στη Δυτική Ευρώπη και στις ανατολικές χώρες, στις χώρες Ανατολικής Ευρώπης, ε, δεν ε, εδρεύει καμία υπηρεσία. Γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό. Ε, είναι τεράστιες αυτές οι διακρίσεις και οι διαφορές. Βλέπω που βρίσκονται όλες οι έδρες. Και βλέπω ότι έχουμε μία από τα ίδια για άλλη μια φορά. Λέμε λοιπόν ότι οι υπηρεσίες πρέπει να βελτιώσουν την ορατότητά τους, δηλαδή να γίνουν πιο προφανείς, πιο εμφανείς στον κόσμο. Ε, ας αλλάξουμε τότε τα πράγματα. Ενώ παραμένουν τα ίδια προβλήματα. Έρχομαι στο θέμα της Ευρωπόλ. Εκεί έχουμε μάθει τα μαθήματά μας. Σε άλλες περιπτώσεις σε αυτή τη διαδικασία έγκρισης της δημοσιονομικής διαχείρισης προσκρούμε στους ίδιους ε, ε, σκοπέλους ξανά και ξανά με την πάραδο των ετών. Εγώ επισκέφτηκα τη Eurofront φέτος. Είδατε πώς ε, χρησιμοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εκεί δουλεύουν σε ένα φανταστικό κάστρο στην Ιρλανδία, δύο βήματα από το Δουβλίνο. Έχετε δει τι εγκαταστάσει τους. Στοιχίζουν πάρα πολλά χρήματα όλα αυτά. Γιατί επενδύουμε συνεχώ σε τέτοιου είδου εγκαταστάσεις και υποδομές. Έχω επισκεφτεί και άλλους οργανισμούς, τις ε, υποδομές που έχουμε στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα. Και τις εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και στην Νεάσο. όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέμε ότι θα έχουμε δεύτερη έδρα. Τι γίνεται με το ενίκιο αυτή τη δεύτερη έδρα. και ω προ τη διαφάνεια τη ΕΑΣΟ, το είπε και ο Συνάδελφο κ. Σαρβάμα, τίθεται πάρα, πολλά, πάρα πολλέ ερωτήσεις. Γιατί θα πρέπει η ΕΑΣΟ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη για το Άσυλο, να προσλαμβάνει προσωπικό μέσω από άλλε υπηρεσίε και διάφορε επιχειρήσει, Γιατί να μπορεί να προσλάβει το δικό τη προσωπικό και να πρέπει να περνάει από ενδιάμεσου και μεσάζοντες. Είναι πολύ θεμητά αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί η κινητικότητα των υπηρεσιών, η γεωγραφική τους κατανομή, γιατί και τα νίκια είναι πανάκριβα εκεί που βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις δεν είναι οι πιο κατάλληλες και ε, γιατί η εργασία την οποία φερούσε πέρα ενδεχομένω επιδέχεται πολλών ε, μικρών ίσως και μεγαλύτερων βελτιώσεων. Από εκεί και πέρα να γίνει καλύτερη επικοινωνία ε, της δουλειάς που κάνουν οι οργανισμοί. Από τη στιγμή που δεν γίνεται καλύτερη η επικοινωνία να μην μας εκπλήσει ότι ο κόσμος απομακρύνεται, οι λαοί απομακρύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν την καταλαβαίνουν. Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μέρη, η Ελλάδα, η Πολωνία, ε, πάρα πολλά κράτη, ενδεχομένω και η Γαλλία, όπου η συνεργασία με αυτές τις χώρες και αυτά τα κράτη σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά περίπλοκοι και πολύ συχνά ενίοτε μάλλον θα έλεγα ότι ακούμε και τελείως παράλογα πράγματα. Μιλούμε για λεπτομέρειες στήριξη σε επίπεδο υποδομών και εγκαταστάσεων που είναι απλά λεπτομερείς και ξαφνικά γίνονται εξαιρετικά περίπλοκες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, η έδρα των οργανισμών είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ασκείται κριτική στο θέμα της συνεργασίας. Θα πρέπει να έχουμε προοπτική. Και αν δούμε το δίκτυο των οργανισμών πριν από τρία χρόνια, ποια εικόνα παρουσίαζε και ποια εικόνα παρουσιάζει σήμερα, βλέπουμε ότι έχουμε προοδεύσει πάρα πολύ. Χρειάζεται όμως περισσότερη πρόοδος. Θα πρέπει να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα και αυτό είναι κάτι που εγώ ε, το αποτιμώ με πολύ θετικό πρόσημο. Να συγχαρούμε τους διευθυντές των υπηρεσιών που έχουν ε, βελτιώσει τους οργανισμούς των οποίων προείστανται. Ζητώ συγγνώμη που ξαναζήτησα το λόγο και ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε που ακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σταθούμε λίγο σε όλα αυτά τα ζητήματα και αν είχαμε και περισσότερους βουλευτές ε, παρόντες, ενδεχομένως θα ήταν και πολύ πιο επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες στον συνάδελφο και Βεβαίως είναι σημαντικές οι υπηρεσίες και οπωσδήποτε ε, θα καταθέσουμε και τις σχετικές τροπολογίες για να δείτε πόσο σημαντικές ε, τις θεωρούμε αλλά όταν υπάρχουν ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα στην Επιτροπή, εγώ τα τηρώ. Και αυτό είναι ε, καμιά φορά ο κίνδυνος όταν πηγαίνει κανείς πολύ γρήγορα, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Όπως και οι άλλες εκθέσεις άλλωστε. Με μεγάλη ευχαρίστηση άκουσα και διάσα την έκθεση του Μπαρτστάς και έχω κάποιες ερωτήσεις. Ναι, ναι. Αρκετέ. Για να ξεκινήσω. Η αυτήν την στιγμή ε, ίσως φαίνεται ότι δεν θα λάβει απαλλαγή γιατί υπάρχουν προβλήματα με την διαχείριση και πρέπει να περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Αλλά εάν δούμε και τις άλλες μεμονωμένες εκθέσεις ε, υπάρχουν διάφορα παραδείγματα. Το Ευρωπαϊκό ε, Ίδρυμα Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Στην πρώτη παράγραφο εκεί πέρα διαβάζουμε ότι ο εισηγητής ανησυχεί για τα ευρήματα του 2012, 2013 και 2015 του ελεγκτικού συνεδρίου και το ότι δεν έχουν υπάρξει ακόμα διορθωτικές δράσεις ε, και επίσης και σε μια άλλη έκθεση διαβάζουμε παρόμοια πράγματα και πραγματικά αναρωτιέμαι ποιο είναι το όριο στο οποίο δίνουμε απαλλαγή όταν εδώ πέρα δεν έχουν ληφθεί κάποιες διορθωτικές ε, δράσεις. Είναι ένα ε, ερώτημα το οποίο βεβαίως ε, αφορά την γενικότερη φιλοσοφία μας. Δεύτερον, η ορατότητα λεγόμενη των υπηρεσιών αυτών. Και εδώ πέρα ένα θέμα της ε, φιλοσοφίας μας. Ε, γιατί ακριβώς ε, λέμε ότι είναι πάρα πολύ γνωστά στα κράτη-μέλη. Αν ρωτήσουμε τους Ολλανδούς που βρίσκεται η Eurojust και το ξέρουν κάνα δύο Ολλανδοί ότι βρίσκεται στην Ολλανδία. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το οποίο λέτε highly visible. Ναι, εσείς το ξέρετε, εντάξει. Το ότι το να είναι έτσι η κατάσταση ε, σε ένα κράτος μέλος. Εντάξει, πόσοι το ξέρουν στη Μάλτα, ας πούμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς η δημοσιότητα. Παραδείγματο χάρη, η υπηρεσία τροφίμων δίνει πιστοποιητικά, η υπηρεσία χημικών δίνει εγκρίσεις και κανείς ε, δεν ξέρει ε, που ε, βρίσκονται. Λοιπόν, δεν είναι θετικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας δημιουργεί μόνιμη ανησυχία, όπως επίσης και το ότι υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες εργάζονται στον ίδιο τομέα και έχουν συνεχώς όλο και περισσότερες επαφές, κάτι που είναι θετικό βεβαίως για τους ίδιους, αλλά είναι δύσκολο για εμάς να εξηγήσουμε το ότι υπάρχει η αστυνομική ακαδημία στην Αυστρία και η Europol ε, στην ε, Χάγη, το οποίο είναι και περίεργο και εμφανίζεται κάθε χρόνο στις παρατηρήσεις της ε, απαλλαγής. Και αυτό θα πρέπει να το δουν ακριβώς ε, αυτοί οι οποίοι ε, χαράζουν την πολιτική. Το Συμβούλιο Υπουργών δηλαδή και η Κομισιόν. Μετά για την χρηματοδότηση είναι θετικό το ότι κάποιες υπηρεσίες έχουν τα δικά τους έξοδα μέσω των τελών που επιβάλλουν, αλλά βλέπουμε ότι δεν πηγαίνουν απευθείας στις υπηρεσίες αυτές, όπως και στο Dieselgate επίσης το ίδιο συνέβη. Περνάνε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτούνται ξανά από τον προϋπολογισμό θα έπρεπε να έχουν μια πιο σταθερή ροή ε, εισοδήματος και να είναι πιο ανεξάρτητη. Επίσης με ανησυχία διάβασα ότι έχουμε ε, εξοικονόμηση στο θέμα του προσωπικού κάτι το οποίο μεταφράζεται σε πρόσληψη εξωτερικών ε, συνεργατών ε, και μια έτσι λεγόμενη δεξαμενή απασχόλησης ε, και κινητικότητας θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες εναλλακτικές και εμείς να σκεφτούμε το τι μπορεί να γίνει. Η κινητικότητα μεταξύ τέτοιων υπηρεσιών βεβαίως είναι ένα περίεργο σύστημα γιατί μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες ειδικότητε και εξειδίκευση και δεν σημαίνει ότι μεταφέρονται αυτομάτως από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Το δίκτυο το επενούμε εδώ πέρα Βεβαίω δεν υπήρχε κάποια συγκεκριμένη και σταθερή δομή τα τελευταία χρόνια αλλά εγώ θα ήθελα να δω κάποια πράγματα περισσότερο για τις αρμοδιότητες αυτού του ε, δικτύου. Εντάξει, είναι αυτόνομες αυτές οι υπηρεσίες, αλλά εντάξει, πέρα από το να τα διευκολύνουμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Μπορεί να είναι παραδείγματο χάρη να, όπως βλέπουμε στους δικαστές οι οποίοι εντάξει είναι ε, ανεξάρτητη, αλλά όσον αφορά την πρακτική οργάνωση της ε, δουλειάς υπάρχουν ε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές και κάποια οργάνωση. Ναι, ναι, έχω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις, οποίες δεν θα κάνω. Θεωρώ ότι το ελεγκτικό συνέδριο τελικά δεν ε, έκανε αρκετούς έλεγχους και θεωρεί ότι δεν έγιναν και αρκετοί αυτοέλεγχοι στα... στις υπηρεσίες αυτές. Και υπάρχει ακριβώς εδώ πέρα και ένας κίνδυνος ε, όσον αφορά την φήμη και την εικόνα αυτών των υπηρεσιών το οποίο οπωσδήποτε θα καταθέσουμε και σε μια τροπολογία και τέλος θα μιλήσουν προσεχώς οι αρχηγοί των κυβερνήσεων για τον προπολογισμό, το πώς θα διαχειριστούν τα χρήματά μας λογικά και θα πρέπει να εξετάσουν. Έχει νόημα, παραδείγματο χάνει η υπηρεσία σιδηροδρόμων να έχει δύο έδρε επειδή κάποτε είχε συμφωνηθεί ότι αυτό ήταν το σωστό. Να πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τα πράγματα λογικά γιατί βεβαίως ε, δεν φταίνε οι ίδιες αλλά οι αποφάσεις ε, του Συμβουλίου. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω θα επανέλθουμε σε κάποια ζητήματα και στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε με την απαλλαγή, Μπάρτ, να σας πω ότι έχουμε εδώ πέρα τον υποδιευθυντή της ε, DigiHome, αρμόδιο για την ΕΑΖΟ, αλλά ε, δεν το απευθύνατε κάποια ερώτηση άμεσα. Αν θέλετε να του δώσουμε τον λόγο, ευχαριστώ. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Νομίζω ότι ο εισηγητής ένα πολύ λεπτό ζήτημα το αντιμετωπίσε με πολύ μεγάλη επιμέλεια και στηρίζω όλες τις προτάσεις και τις συστάσεις του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπάρτ, παρακαλώ, έχετε το λόγο είστε εισηγητής για να βγάλετε τα τελικά συμπεράσματα. ευχαριστώ Μαρτίνα, ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις θετικές παρατηρήσεις να αναφερθώ λίγο σε κάποιες παρατηρήσεις ιδιαίτερος του Ντένις. Ε, υπήρξε νομίζω μια παρατήρηση για την έκθεση του Όλαφ ε, για την ΕΑΖΟ και για το τέλος του καλοκαιριού. Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου περιμένουμε επισήμως ε, έχω άτυπες επαφές με τον Όλαφ, αλλά γνωρίζω μόνο το ότι εργάζονται εντατικά πάνω στο θέμα και ότι κανονικά θα πρέπει να αναβληθεί η αναλογή του ΕΑΖΟ και μπορούμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη και τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου οπότε κανονικά θα γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την έρευνα. Εν πάση περιπτώσει αν αναβάλουμε αυτήν την απαλλαγή και ξεκινήσουμε μέσα Σεπτεμβρίου νομίζω ότι θα έχουμε επαφές με τον Όλαφ για να ξέρουμε εάν τα πράγματα ε, μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε ή όχι και πιθανώς να μην ε, δώσουμε απαλλαγή. Ε, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον τρόπο να πιέσουμε τον Όλαφ να σεβαστεί κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να το δούμε με τον Διευθυντή για να πάνε να κυλήσουν τα πράγματα σωστά. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, να αφαιρθώ σε αυτά τα οποία είπα τώρα. Ναι, υπάρχει μια ανισορροπία, θα έλεγα, γιατί υπάρχει αναβολή για την ΕΑΖΟ, ενώ στα άλλα έχουμε κάποιες σταθερές ε, θα έλεγα παρατηρήσεις εντάξει το αντιλαμβάνομαι είναι μια σωστή παρατήρηση θα έλεγα ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε πράγματι με τους χειοδησηγητές δηλαδή ποιο είναι το όριο όπως είπατε και εσείς το όριο εγώ θα έλεγα ότι είναι η έρευνα του Όλαφ αυτό είναι το θέμα τα υπόλοιπα εντάξει υπάρχουν επιφυλάξεις, ε, αλλά και οι ομάδες ε, θα έλεγα ότι ήταν υπέρ ε, κατά πλειοψηφία του να δοθεί απαλλαγή στις άλλες περιπτώσεις. Και είπαμε ακριβώ να τα δούμε όλα αυτά και στις τροπολογίες όταν θα κατατεθούν ε, τον Μάρτιο. Σε ευχαριστώ λοιπόν Ντένις για αυτήν την παρατήρηση. Δεύτερον, για την δημοσιότητα των υπηρεσιών αυτών. Τι εννοώ εδώ πέρα. Ε, δεν εννοώ απαραίτητα. Ναι, ίσως να μην ήταν ε, τόσο καλή η διατύπωση. Εννοώ ότι είναι ιδιαίτερος μεγάλη σε σχέση με τους ανθρώπους, ε, τις οργανώσεις εκείνες οι οποίες έχουν κάποια επαφή με το έργο των υπηρεσιών αυτών. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική του ασύλου γνωρίζουν το τι κάνει η Άζο, ε, τι κάνει η Frontex. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ασφάλεια τροφίμων γνωρίζουν το τι κάνει η ΕΦΣΑ και τις σχετικές συζητήσεις. Το ίδιο και με την υπηρεσία φαρμάκων. Δηλαδή, οι ομάδες στόχοι που έχουν σχέση με το έργο αυτών των υπηρεσιών τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία σε δέσμες ε, μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών, Frontex, EASO, Europol κτλ. Αναφέρατε και εσείς και την Αστυνομική Ακαδημία που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Πράγματι είναι μια συζήτηση αυτή. Η όλη συζήτηση πράγματι για παραδείγματος χάρη το τι γίνεται με την ΕΦΣΑ όπου πρέπει να υπάρχει όπως είπε και ο Ντένις μια ε, ξεκάθαρη γραμμή όταν μιλάμε για την πληρωμή των τελών ε, ε, όταν κάποιος πληρώνει τέλη σημαίνει ότι έχει την απέτηση ο φακελός του να τύχει της ανάλογης προσοχή Βεβαίω μετά αυτά τα τέλη πηγαίνουν στην Κομισιόν για να ξανααποδοθούν στο, στην ε, εκάστοτε υπηρεσία και αυτό είναι ένα ζήτημα. Επίσης ε, σημαντικό θέμα είναι ακριβώ ε, το θέμα της οικονομίας στο προσωπικό κανόνα κανόνας του 5% ακούστηκε και στις ακροάσεις όταν είχαν έρθει οι αποκεντρωμένες αυτές τι υπηρεσίες εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο και όπως είπαμε αυτό οδήγησε σε υπερβολική πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών που δικαίως βεβαίως μας ανησυχεί. Το γεγονό ότι μιλάμε για ένα δίκτυο επίσης για συνεργασία, για συντονισμό εντάξει, ίσως πρέπει να καθοριστεί καλύτερα σε μια παράγραφο στην οριζόντια έκθεση το ποιε είναι οι αρμοδιότητε αυτού του δικτύου. Νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει πολύ στις ε, περαιτέρω συζητήσεις και ίσως αυτό αποτελεί και ένα επιχείρημα για να πείσουμε και το Συμβούλιο, το οποίο ήταν πολύ επιφυλακτικό. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό πράγματι έχετε απολύτως ε, δίκαιο εδώ και Δεν μπορώ να, δεν μπορώ να διαβάσω τα γραμματά μου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάτι ακόμα. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Εύσα που κάνει τον συντονισμό και το έκανε με τρόπο υποδειγματικό. Οπωσδήποτε ο Έρολ ε, εκεί πέρα στην Ηλιόλου, στη έδρα του, στην ε, Πάρμα κάνει καλή δουλειά και να ευχαριστήσω και όσους με βοήθησαν, την ε, Σεσίλ που κάθεται εκεί και ήταν ε, πραγματικά πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της και μπήκε στη δουλειά εκεί πέρα σαν Pitbull και καθοδήγησε μένα και τον Ροκ Χαρόμπι και τον Ρόμπερτο Χοντίνα τους ε, δύο συμβούλους ε, των Πρασίνων μας είπαν πρέπει να σεβαστείτε, μας είπε πρέπει να σεβαστείτε αυτό, αυτό, πότε θα αντιδράσουν, τι απαντήσεις θα σας δώσουν και ήταν πραγματικά πολύ αποτελεσματική ε, και κατάφερε να γίνουν όλα εγκαίρως. Ήταν η πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε. Ήταν νομίζω και η πρώτη μεγάλη τέτοια δουλειά που είχα αναλάβει. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ και τους Ρόκου και Ρόμπερτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπάρτ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Πρόεδρο, να σας πω ότι όλοι διαμαρτυρήθηκαν για την ισχνή συμμετοχή για το ότι η συνεδρίαση προβλέπεται στις, ε, τη Δευτέρα το απόγευμα. Ίσως πρέπει να αλλάξει αυτό για να έχουμε περισσότερους παρόντες. Και υπάρχει και το θέμα της ε, ε, ε, ισορροπίας της εκπροσώπησης των φίλων, όπως είπε και ο Μπάρτε. Πρέπει να σας πω ότι η ισορροπία στην εκπροσώπηση των φίλων στο Προεδρείο είναι εξαιρετική σήμερα και σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Ναι, πάντα τα καλά γίνονται πριν έρθω. Λοιπόν, ήμουνα σε μια εκδήλωση του κ. Ταγιάννη για έναν Ιταλό συγγραφέα και ξαναρχόμαι, έχουμε την ομάδα εργασίας βέβαια για τις υπηρεσίες. Είχα την προηγουμένη φορά την ευκαιρία να συμμετάσχω. Τώρα δεν πήγα γιατί θεώρησα ότι έχω καλύτερα πράγματα να κάνω. Και έτσι πρώτη ερώτηση. κύριος Δε Ιόγκ, που είναι μέλος, πιστεύει ότι μπορεί να έχει κάποια διαφορετική μοίρα αυτή η ομάδα εργασίας από ό,τι προηγούμενες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα δύσκολο θέμα γιατί ξεκίνησα με μεγάλο ενθουσιασμό ως μέλος της Επιτροπή Διοργανικής Συνεργασίας. Είχαμε μεγάλες ε, προσδοκίες και καταλήξαμε σε κάποια ουσιαστικά σημεία στα οποία είπαμε ναι, καλό είναι η Κομισιόν να ξαναδεί αυτά τα ζητήματα στις ε, πενταετής αξιολογήσεις. Ε, δεν ξέρω τώρα αν ήταν αναγκαία αυτή η δουλειά. Έγιναν κάποιες συζητήσεις οι οποίες οπωσδήποτε ήταν απαραίτητες. Ε, η προσωπική μου αντίληψη ήταν ότι είχαμε μια ευκαιρία για να δούμε το τι θα κάνει η Κομισιόν ε, και με εκθέσεις οι οποίες ε, θα υποβληθούν φέτος και έχουμε πράγματα όπως ε, τα αποτελέσματα των περικοπών του προσωπικού το πιο σαφές αλλά βεβαίως η εντολή θα έλεγα αυτή της ομάδας εργασίας ήταν ε, να καταλήξει σε κάποιες συστάσεις ε, να δούμε παραδείγματος χάρη την ε, συσσωμάτωση να αναγραφούν σε δέσμες κάποιες υπηρεσίες παραδείγματος χάρη οι οποίες έχουν παραπλησίες εντολές στην δουλειά τους και εκεί πέρα μετά σταματάνε τα πράγματα. Και... Βεβαίως, κανείς δεν θέλει να ανοίξει στα αλήθεια αυτό το κουτί της ε, Πανδώρας ε, και βλέπουμε ότι η Κομισιόν μετά θα κάνει την επόμενη έκθεση ε, προόδου όπου τα πραγματικά δύσκολα ζητήματα θα μείνουν κατά μέρος. ή αυτά τα οποία ανέφερε στην προηγούμενη συζήτηση ο Μπαρτ Στάς, παραδείγματος χάρη, όλες οι σχετικές υπηρεσίες με τη δικαιοσύνη να πάνε σε ένα μέρος. Μα αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσει κάπου και η υπηρεσία σύλλου. Αλλά βεβαίως από την άλλη θα αντιδράσει πολύ μάλτα Και έτσι πάνε τα πράγματα στο Συμβούλιο. Το αν έχουν λοιπόν οι ηγέτες ε, το θάρρος να κάνουν κάτι τέτοιο δεν το νομίζω. Είμαι απεσιόδοξο Το έχουμε μετά συγκεκριμένες συζητήσεις που πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστούν ε, γιατί είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για την χρηματοδότηση και την στελέχωση των ε, υπηρεσιών αυτών. Αφενός Μιλήσαμε για τα τέλη τα οποία επιβάλλουν, μιλήσαμε επίσης για το ότι θα πρέπει όταν δεν έχει τέτοια δυνατότητα εμείς ως αρχή προϋπολογισμού να ενισχύσουμε μία τέτοια υπηρεσία και βέβαια να αυξηθεί ταυτόχρονα η λογοδοσία και η ευθύνη και για να αποφευχθεί ακριβώς όπως σας είπα ο κίνδυνος ε, για την φήμη και θα πρέπει να δούμε πως επιβληθούν κάποια επιπλέον κριτήρια γιατί οπωσδήποτε θα μας αποσχολήσει αυτό το θέμα στο μέλλον. Επίσης αυτό το οποίο μόλις ακούσαμε για την εξάρτηση ε, από τα τέλη, το τι πρέπει να γίνεται αν πρέπει να πηγαίνουν απευθεία ή μέσω του προϋπολογισμού της ε, Κομισιόν, αλλά προσωπικά απογοητευτικό ήταν το εξής ε, είδαμε το θέμα της ΕΑΖΑ που υπήρχε ένα πιλωτικό έργο για την ασφάλεια των αεροπλάνων και εκεί πέρα η Κομισιόν υπέβαλε κάποιους δίκτες ε, και το ερώτημα ήταν ποιοι ήταν οι ποιοτικοί ε, δείκτες ε, γιατί ετέθηκε το ζήτημα βεβαίως του ε, τι πληρώνει κάποιος όταν πληρώνει κάποιος τέλει και βεβαίως σε συγκεκριμένη περίπτωση είπαμε ότι θα πρέπει να είναι παραδείγματο χάρη να εξυπηρετεί τον κλάδο εγκαίρος και να είναι φιλικός προς τους συγκεκριμένους ε, πελάτες κτλ. Είναι αυτό ή πρέπει ε, να φροντίζει να είναι όντως ασφαλή τα αεροπλάνα. Και το είχαμε συζητήσει αυτό τότε με την Αντιπρόεδρο Γεωργίευα και τελικά ποτέ δεν λάβαμε κάποια απάντηση σε αυτό το ερώτημα από την ε, Κομισιόν. Είναι λοιπόν αυτό ένα πιλωτικό έργο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί ως υπόδειγμα και από τις άλλες ε, υπηρεσίες. Είναι λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα, Είχε δίκιο η πρόεδρος πράγματι ε, είχαμε πολλές ε, συνεδριάσεις τελικά όμως αναμένουμε να, το τι θα κάνει η Κομισιόν κάτι το οποίο είναι πράγματι Κρίμα. Και ως ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού βεβαίω και εμείς συζητάμε να γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά στον εκάστοτε τομέα. Ναι, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Ντεϊόγκ. Είναι πολλή δουλειά και το είδα και εγώ ίδια. Και πρέπει να ευχαριστούμε τις υπηρεσίες τένισαν τις υπηρεσίες από πάνω ως κάτω οριζόντια κάθετα και διαγώνια και έχουν ε, παράγει πολύ καλό προϊόν, υλικό. Γιατί διαπιστώνεται ότι υπάρχουν υπηρεσίε οι οποίε είναι ανέκανε ακόμα και τα πιο βασικά πράγματα να αποφασίσουν, όπω παραδείγματι τη συγχώνευση υπηρεσιών που είναι κοινέ. Ε, και άρα είναι αδιανόητο το ότι μπορούμε όλα αυτά να τα ξέρουμε αλλά να μην μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση. Και είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητηθεί με το Συμβούλιο, με την Ισπανική Προεδρία. Που χρειάστηκε να το συζητήσω. Είναι ένα θέμα μεγάλο, πολύ ενδιαφέρον για την Επιτροπή των Ελέγχου του Προϋπολογισμού για τον προπολογισμό, πρέπει να το παρακολουθήσουμε όλοι με ενδιαφέρον και είναι προφανές ότι τροφοδοτείται και ο το αντιευρωπαϊκό μένος όταν δεν είμαστε σε θέση εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό, να το έχουμε στην επικαιρότητα, στην ημερήσια μας διάταξη και να κοιτούμε την ε, διαρκή παρουσία των υπηρεσιών στις συζητήσεις. Κρίμα που δεν έχουμε τους εταίρους που θα χρειαζόμασταν στις διαδικασίες αυτές. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ατελείωτη ιστορία λοιπόν. Τι ωραία που ήταν όλα αυτά. Αν θέλει κάποιος το λόγο... Ιδάλλως τα σημειώνουμε. Είδαμε και την επιστολή του Προέδρου. Ναι, εδώ είναι το μόνο που μένει να δούμε τι θα την κάνουμε. Να απαντήσουμε κι εμείς. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις κάποια ιδέα. Τι να κάνουμε με τις συστάσεις αυτές, τις recommendations. Για να υπογραμμίσουμε τη σημασία τους, έχεις κάποια ιδέα, μια επιστολή ενδεχομένως, κάποια άλλη απάντηση προς τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο. Ναι. Θεωρώ ότι η ομάδα εργασία συμφώνησε για τον Ιούλιο φέτος και με τους συντονιστές είπαμε να συντάξουμε μια επιστολή για το τι ακριβώς ε, αναμένουμε γιατί θα πρέπει να καθοριστούν κάποιες ε, προτεραιότητες ε, που θα μπουν μετά σε αυτήν την επιστολή. Νομίζω ότι είναι το πιο αποτελεσματικό αυτό και το συνδέσουμε με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και νομίζω θα μπορούσε ακριβώς να θα υπάρξει αυτή η νέα διάσταση. Την Κομισιόν, την Γενική Γραμματεία, η κυρία Μιχαήλωβα. Um, Ευχαριστώ. Είμαι διαθέσιμη να απαντήσω σε ερωτήσεις σας, αλλά δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη με τη δουλειά των τριών θεσμικών οργάνων Χαιρόμαστε διότι το Κοινοβούλιο έχει στηρίξει τις συστάσεις και εμείς ε, πράττουμε το ίδιο και ενθαρρύνουμε το Συμβούλιο να πράξει και αυτό το ίδιο το συντομότερο δυνατό. Αν έχετε ρωτήσει τη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ναι, το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται, πώς πρέπει να περιμένουμε την εφαρμογή των συστάσεων με τη ε, χρονική απόσταση. Κοιτάξτε. Οι συστάσεις δεν προβλέπω συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα, απευθύνονται στα τρία θεσμικά όργανα, αλλά βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλει αναφορά για όλες τις διαδικασίες, για τη διαδικασία του προπολογισμού και θα διενεργήσει τη δουλειά της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών της. Αλλά δεν έχει ε, καθοριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από καμία σύσταση Όμω τον Ιούλιο είναι η επόμενη συνεδρία των εμπειρογνωμόνων και τα τρία θεσμικά όργανα υποτίθεται ότι θα ξανασυναντηθούν, θα κάνουν τον απολογισμό τη ε, κατάσταση και θα αναφέρουν την επίδευξη πρόοδου. Θα μπορούσε αυτό να είναι η πρώτη ευκαιρία, έτσι δεν είναι. Ναι, εξαιρετικό. Αν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα δεν μα εμποδίζει και τίποτα να ξεκινήσουμε αμέσω. Και αύριο δηλαδή. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν περνούμε στην υλοποίηση. χωρί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να μου το εξηγήσετε λίγο. Ναι, η ομάδα της στην τελευταία συνεδρίαση συμφώνησε ότι κάθε θεσμικό όργανο θα ακολουθήσει τη δική του εσωτερική διαδικασία για να στηρίξει αυτές τις συστάσεις. Και άπαξ ε, τις, τις στηρίξουν και τα τρία θεσμικά όργανα, μπορεί η διαθεσμική και διοργανική ομάδα εργασίας να συνεχίσει, να πάρει τη σκητάλη. Το Συμβούλιο δεν το έχει κάνει ακόμα, δεν έχει ολοκληρώσει δηλαδή, τη δική του εσωτερική διαδικασία. Αυτό περιμένουμε. Ωραία, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να αρχίσουμε σαν τις μελισσούλες να ζουνίζουμε γεμάτη επιμέλεια και διάθεση για δουλειά. Ποιος θα τα αποφασίσει όλα αυτά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ε, περιμένουμε δέκα χρόνια τώρα. Θέλω ένα χρονοδιάγραμμα που θα μου λέει μέχρι εκείνο το σημείο θα έχετε τεθεί σε εφαρμογή. Μπορείτε. Να σας πω για άλλη μια φορά ότι καμία από τις συστάσεις δεν προβλέπει συγκεκριμένη υποχρέωση για ε, τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος και η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να τηρεί ενήμερους τους πάντες για τη διαδικασία. Οι συστάσεις έχουν εγκριθεί από τα έχουν συμφωνηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα και πρέπει να εγκριθούν επισήμω με την εσωτερική διαδικασία του κάθε θεσμικού οργάνου. Ακριβώς. Οι συστάσεις, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Συγχωνεύσεις, κλεισίματα, μεταβίβαση καθηκόντων. Χωρίς να λέει ακριβώς κάντε το, αλλά δείχνει τι μπορεί κανείς να κάνει αν θέλει να κάνει κάτι. Άρα πιστεύουμε ότι θα πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συνεχίσει να δουλεύει πάνω στο θέμα αυτό και να κάνει προτάσεις. Υπάρχει όμως αυτή η βούληση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο. Να κοιτάει ο ένα τον άλλον συνέχεια και να περιμένει ποιο θα κινείται πρώτο. Είναι καθήκον τη Επιτροπή να προωθήσει την υπόθεση αυτή. Πρέπει να διατυπώσει προτάσει. Άλλων δεν έχουν γίνει δεκτές άλλη ιστορία, άλλον θα κατηγορούμε. Αλλά το να καθόμαστε και να περιμένουμε δεν είναι καλή ιδέα. Ναι, οι συστάσεις είναι, έχουν συνταχθεί με τρόπο κατά τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τους τις εσωτερικές διαδικασίες κάθε οργάνου η Επιτροπή δουλεύει με βάση την εσωτερική της διαδικασία. Αν προκύψουν νομοθετικές προτάσεις, βεβαίως ε, η Επιτροπή έχει την ευθύνη και την υποχρέωση να τις ε, παρουσιάσει και να τις προωθήσει. Καλώ λοιπόν, Τένις. Ε, τον Ιούλιο έχουμε αυτή την πρώτη ομάδα εργασία. Άρα, μετά την πρώτη συνεδρίαση, μπορούμε να κοιτάξουμε, να δώσουμε λίγο χρόνο, να συζητήσουμε και να πούμε αυτά είναι τα επόμενα βήματα. Γι' αυτό παρακαλώ την Επιτροπή να μα έχει έτοιμα μέχρι το Σεπτέμβριο τα πρώτα βήματα για να κλείσει αυτό το θέμα πια. Φτάνει, ε, μπορούμε. Παρακαλώ. Ναι. Αλλά για προς υπεράσπιση της ε, Κομισιόν θα πρέπει να πούμε πως ε, θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία αυτά πριν από την συνεδρίαση του Ιουλίου του 2018 για να δούμε ε, βεβαίω αν ε, συμφωνούμε και με τις ε, συστάσεις. Τα είχαμε συμφωνήσει αυτά στην ομάδα εργασίας μεταξύ μας πριν από μισό έτος και τα πράγματα τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα ως υλικό που θα πρέπει να μας προμηθεύσει η Κομισιόν καλό είναι να μην περιμένουμε μέχρι τον Ιούλιο να έρθουν αλλά να έρθουν κάπου λίγο πιο νωρί ε, Τα είχαμε πει αυτά και με τον Γιάννη Γκάιερ από την Επιτροπή Προπολογισμού. Νομίζω θα είναι μια καλή αρχή. Ωραία λοιπόν, τότε να προσπαθήσουμε να το πείσουμε για το Μάιο μια ε, ημερομηνία που θα προσκαλέσουμε την ε, κυρία από την Γενική Γραμματεία και μετά πάλι θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, λοιπόν, το Μάιο, η υλοποίηση συστάσεων και προσδιορισμός των προσεχών βημάτων με στενή παρακολούθηση. Αλλά βέβαια ξέρετε ότι όταν προσκαλούμε τους επικεφαλείς των υπηρεσιών είναι κακό. Για να δούμε αν θα βρει το δρόμο και ο Γενικός Γραμματέας της Επιτροπής. Ωραία, κλείνουμε το θέμα αυτό της ημερήσης διάταξης. Κύριε Σέις θα μας κάνει την παρουσίαση του θέματος του, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις πριν προβώ σε ορισμένα σχόλια για τις κοινέ επιχειρήσεις τις οποίες συζητούμε ε, για φέτος, τα joint undertakings. Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε μια πολύ σημαντική έκθεση που προέκυψε από το ελεγκτικό συνέδριο και η οποία δημοσιεύεται άπαξ ετησίως. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, απεικονίσουμε σωστά ε, τα πορίσματα αυτών των εκθέσεων ε, του ελεκτικού συνεδρίου αλλά και τα πορίσματα των συζητήσεων στις ακροάσεις που έχουμε εμείς κάνει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σκοπός είναι να παρουσιάσουμε και τα καλά και τα κακά να αποδώσουμε μια δίκαιη εικόνα για τις κοινέ επιχειρήσεις και να μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι στο στόχαστρο της αρνητικής άποψης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άλλωστε, εγώ προτείνω να εγκρίνουμε την απαλλαγή στη δημοσιονομική διαχείριση για όλες τις κοινέ επιχειρήσεις και το λέω αυτό ευθύ εξ αρχής, να μην νιώσει κανείς ότι βρίσκεται στο εδόλιο. Ωστόσο, πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την έρευνα, για την καινοτομία, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτές οι κοινέ επιχειρήσεις σχετίζονται άμεσα με όλα αυτά. Και αν δούμε το έτος 2016, μιλούμε για 1,8 δις ευρώ. Είναι μια πολύ ε, πλούσια εταιρική σχέση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι δαπάνε του δημοσίου τομέα από το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να απεικονίζονται με τρόπο κατά τον οποίο θα υπάρχει απόλυτη λόγοδοσία ε, και με βάση τα προκρινόμενα από το ελεκτικό συνέδριο. Επομένως, εμείς θέλουμε να ρίξουμε φως στα καλά αποτελέσματα, να τα αναδείξουμε, να πούμε σαφήνεια τι είναι αυτό το οποίο δουλεύει και θέλουμε με εξίσου μεγάλη σαφήνεια να πούμε ποιο είναι αυτό το οποίο πράγματι πρέπει να βελτιωθεί και μπορεί να βελτιωθεί με δεδομένο το βελινεκές του προϋπολογισμού. Μιλάμε για 1,8 δίσο ευρώ, σχεδόν το 3% ίσως του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Έχουμε το Shift to Rail, το Excel και το EMI. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και γι' αυτό θα ήθελα να σταθώ σε κάθε μία, σε κάθε μία από αυτές τις κοινοπραξίες ή κοινέ επιχειρήσεις και να μιλήσω ε, για τα πορίσματά μας. Μιλούμε για εσωτερικά συστήματα ελέγχου και τονίζουμε αυτά τα οποία μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον. Ίσως κάποιοι θα απογοητευθούν και θα ανησυχήσουν για τη διατύπωση που έχω βάλει στην έκθεσή μου, αλλά τη στηρίζω και επιμένω, γιατί είναι σημαντική και πρέπει να μιλήσουμε με απλά λόγια και να μιλήσουμε απλά για το τι όντως δουλεύει και για το τι όντως δεν δουλεύει. Δεν είναι φρικτή κριτική είναι απόπειρα και προσπάθεια να έχουμε βελτιώσει στα συστήματα ελέγχου για το μέλλον, γιατί είναι πολλά τα χρήματα που υπησέρχονται εδώ. Επομένως, έχετε την έκθεσή μου, θα υποβάλω και επιπρόσθετες τροπολογίες για σφάλματα που ενδεχομένω έχουν γίνει στην αρχική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για πράγματα που έχουν έλθει στο φως και έχουν προκύψει ενδιαμέσως και έκτοτε ε, ε, από τις ακροάσεις και μετά. Όμως για τα καινοτόμα φάρμακα, για παράδειγμα, για την κοινή επιχείρηση πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα, το ΙΜΗ, Είπαμε ότι τρία, είναι η τρίτη χρονιά που είμαστε κάτω από το κατόφλι του 75% για για τις πιστώσεις στο προϋπολογισμό appropriations και η συνεισφορά του κλάδου πρέπει να αξιολογηθεί επιτέλους και να δούμε κατά πόσο φτάνει σε αυτό το οποίο περιμέναμε. Και λέμε ότι είναι πολύ σημαντική η καθυστέρηση στις πληρωμές σε βασικούς πελάτες όπως είναι τα πανεπιστήμια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό πλήττει ιδιαίτερο στη δυνατότητά τους για έρευνα και καινοτομία και Είχα κάποιες εξηγήσει, μου είπαν οι συνομιλητές κάποιοι λόγοι, ε, για κάποιους λόγους που εξηγούν αυτές τις καθυστερήσεις και άρα θα υποβάλω τροπολογίες για να ε, ε, υπάρξουν αυτές οι αιτιολογήσεις για το Excel, κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία. Πρέπει να σας πω ότι 24 κράτη έχουν κάνει συνεισφορές το 2016, 4,9% του συνόλου των συνεισφορών Άρα προσπαθούμε να προσελκύσουμε την προσοχή των κρατών που συμμετέχουν να συμβάλλουν περισσότερο για να μην μπει στο πάγο αυτό και να φέρει αποτελέσματα. Για το shift to rail, ε, μεταστροφή προς το σιδηρόδρομο, ήταν η πρώτη χρονιά. Έχω πολλές ανησυχίες για τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στα θέματα αυτά τα shift to rail και να αναγνωρίσω και την πρόοδο που έχει γίνει Τώρα, Fusion for Energy, συγχώνευση για την ενέργεια. Είναι ένα πολύ σημαντικό project αυτό. Η καθυστέρηση είναι 15 ετών. Καταλαβαίνω τη λογική, τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, αλλά πρέπει να το πούμε, πρέπει να την αναφέρουμε γιατί θα ε, χρειαστεί τεράστια συνεισφορά στο μέλλον για να μην καθυστερήσει το πρόγραμμα. Υπάρχει το κόστος αφοπλισμού. Αυτό ακούστηκε στην ακρόαση και θα υποβάλω τροπολογίες για να ε, συμπεριλάβω τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακρόαση. Αλλά χαίρομαι για τη στρατηγική που υιοθετήθηκε το 2016. Για το Sea Survey 1,7 δις είναι οι συνεισφορές σε ρευστό που αναμένοντας στα τέλη του 2016 δεν είχε γίνει καμία συνεισφορά. Είμαστε σε αρχικό στάδιο. Το παρακολουθούμε εκ του συνεγγύς για το ΣΕΣΑΡ, Κοινή Επιχείρηση Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, για το Clean Sky, την ε, αεροναυτική και το περιβάλλον. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συνεισφορές 800 εκατομμυρίων ευρώ όμως έχουν, γίνει μόνο, έχουν δοθεί μόνο τα μισά για τη συγκεκριμένη οικονομική χρήση και για την κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων διάφορα μέλη της ε, κοινοπραξίας αυτής είπαν ότι ήδη τους λογαριασμοί για τη χρήση 2016 δεν είχαν κλείσει, επομένως δεν μπορούν να συνεισφέρουν με συγκεκριμένα στοιχεία και τα στοιχεία δεν είναι ακριβή. Άρα, στις εκθέσεις λοιπόν αυτές τονίζουμε και αυτά που πρέπει να βελτιωθούν αλλά και αυτά που πραγματικά είναι σημαντικά και που έχουν γίνει ήδη βελτιώσεις. Προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά, τις θετικές και αρνητικές ε, διατυπώσεις. Επαναλαμβάνω, δεν προτείνω να μην εγκρίνουμε την απαλλαγή. Προτείνω να εγκρίνουμε την απαλλαγή ε, για τη δημοσιονομική διαχείριση. Ωστόσο, ε, εκεί όπου πρέπει να γίνουν βελτιώσεις, να τις τονίσουμε για να γίνουν και μπορούν να γίνουν και περιμένω να υποβάλω και εγώ νέες τροπολογίες αλλά και εσείς για να συμπεριλάβουμε τα νέα στοιχεία που προέκυψαν ε, ε, μετά από τις ακροάσεις και έτσι να είναι πιο εμπεριστατωμένη η έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ κύριο Σαγουάρμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά ε, σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Χέις, είναι εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ε, διατύπωση ξεκάθαρη. Και χαίρομαι που ο προηγούμενος ομιλητής το τόνισε αυτό. Δεν πρέπει κανείς να θεωρήσει ότι είναι άδικη κριτική που στρέφεται εναντίον του ιδίου. Αντιθέτως, αυτό είναι ο πυρήνας της δουλειάς μας όσο ευρωβουλευτές που ασχολούμαστε με την απαλλαγή, που εγκρίνουμε την απαλλαγή για τη δημοσιονομική διαχείριση ή μη. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Και νομίζω ότι η δουλειά που έχει γίνει είναι εξαιρετική. Ε, και εδώ πρέπει κανείς να είναι πολύ ειλικρινής και πολύ σαφής για να ακουστεί η άποψή του και να γίνει αντιληπτή και από τους οργανισμούς, τις επιχειρίες, τις ε, ε, υπηρεσίες, τις κοινέ επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, ε, είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία αυτή, μια διαβίου διαδικασία αν θέλετε, ε, έτσι ώστε όλα, όλοι αυτοί οι φορείς, όλες αυτές οι υπηρεσίες, όλα αυτά τα όργανα, όποια ε, μορφή και αν έχουν, να λειτουργήσουν καλύτερα από τη στιγμή που χρηματοδοτούνται με τα χρήματα των φορολογουμένων. Επί της ουσίας, ε, με ικανοποίηση σημειώνω ότι δίδεται πολύ προσοχή στις συνεισφορές και αυτό είναι πράγματι κάτι το πολύ σημαντικό. Και για το θέμα του ΙΤΕΡ, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύνδεξης, είναι κάτι που το έχουμε από πάντα, αλλά ε, πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί και ακριβείς, να ε, ουρλιάξουμε Ξέρουμε όλοι ότι αυτοί εκεί ε, κάνουν το ό,τι καλύτερο μπορούν. Όμως είναι μια πολύ σημαντική επιχείρηση και άρα ο ρόλος μας ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα δώσουμε την απαλλαγή είναι ακόμα πιο σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ. Πώς... Πρόεδρε, ευχαριστώ και καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ τον συνάδελφο κύριο Χέις για την καλή προετοιμασία των εκθέσεων για την, ε, που παρουσιάζουν τις ικανοποιητικά, πολύ ικανοποιητικά τις εξελίξεις στις κοινέ επιχειρήσεις, οι κοινοπραξίε. Λίγες τροπολογίες έχω να καταθέσω τεχνικού χαρακτήρα και ξεκινώ με το ΙΤΕΡ που επί το πλήστον συζητούμε, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους στο σύνολο. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου έχει μια παραπλανητική δήλωση, ότι δηλαδή δεν έχουν υπολογιστεί συνολικά οι δαπάνες. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. έχουν προβλεφθεί σε συνεργασία και με την ε, Γαλλία χώρα υποδοχή στα 530 εκατομμύρια για την ενεργοποίηση επειδή δεν έχει προσδιοριστεί χρονοδιάγραμμα και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ποιος είναι ο εταίρος για να γίνει η συμφωνία, εκεί λείπει η τελική αξιολόγηση του κόστους. Ένα άλλο σημείο Το οποίο διαφώνησα με τον ε, εισηγητή ήταν μια κάπως αποστασιοποιημένη δήλωση σε σχέση με τις συνέπειες του Brexit. Εγώ βλέπω ότι η Βρετανία ενδιαφέρεται και με Twitter αλλά και με το γενικότερο τομέα της έρευνας της σύνδεξης να διατηρήσει στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ είναι σαφώς ε, άνισος ο επιμερισμός των, ε, της συμμετοχής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιδιωτικού τομέα. Ενώ οι πληρωμές λοιπόν είναι από τον 2020 και τα σχετικά έργα ως προσωρινές πληρωμές, η επιχειρήσεις καταβάλουν τα ποσά με την ολοκλήρωση των έργων και μόνο και μάλιστα μετά την πρώτη φάση λειτουργίας. Και οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τηρήσουν τις αρχές της αναλογικότητας, την αρχή της αναλογικότητας στην διαχείριση. Έτσι λοιπόν, θα ήταν καλό να είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα τα προγράμματα αυτά του όρου 2020. Είναι ένα εργαλείο καλό, είναι μια κοινοπραξία γερή, είναι καλό να την υποστηρίξουμε. Υπάρχουν ωστόσο συνδεδεμένα προβλήματα, κίνδυνοι, οικονομικοί, δημοσιονομικοί και σε αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειάζεται δηλαδή μια τακτοποίηση, χρειάζεται τακτική μηχανισμοί δημοσιονομικού ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και την κατάλληλη χρήση των μηχανισμών αυτών. Και γι' αυτό πάνω από όλα πρέπει να επενούμε τις κοινοπραξίες αυτές, τις κοινέ επιχειρήσεις, όχι να τις ε, κατακρίνουμε. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή ότι πρέπει να ενισχύσουμε την επικοινωνιακή διάσταση. Πρέπει εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα να συμμετέχουν περισσότερο και να υπάρχει καλύτερη ε, επικοινωνία με την κοινή γνώμη, καλύτερη κοινοποίηση δηλαδή. Καλώς, ε, έχω μια ερώτηση για την έκθεση 6,6 δις ήτρε, ήτερ, μάλλον. Και εμφανίζονται και 4 δις θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσει λίγο η Επιτροπή τι είναι αυτά τα χρήματα ή το ίτερ, DG είναι. Γιατί θα είμαι αρκετέ ε, συνεδριάσεις με τους υπεύθυνους ίτερ. Μας έλεγαν ότι είναι τα τελευταία, τα αξιόπιστα νούμερα, τα 6,6 αυτά δις. Αλλά αν βλέπουμε ένα πρόσθετο ποσό, άλλα 4 δις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρήσουμε και πολύ αξιόπιστα αυτά που μας είχατε πει. Παρακαλώ. Move, Γκάριμπα, ο Βάσιλε, Connect, η Μπέρνες, Νόρστετ, εμεί. Για να δούμε ο κύριος Γκάριμπα πρώτος και τυχερός. Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Αίσερ, τον εισηγητή για την έκθεσή του. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που ακούμε την ε, πρότασή του για την έγκριση της απαλλαγής για ε, το ΙΤΕΡ, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύνδεξης. Πράγματι, η έκθεση είναι σωστή και οι συνάδελφοι αλλά και ο ίδιος ο θα υποβάλει τροπολογίες από ό,τι έχω καταλάβω για να διευκρινίσει κάποια ε, σημεία της έκθεσης που χρήζουν διευκρινήσεων, ε, για παράδειγμα στα εδάφια που αναφέρονται στην Επιτροπή. Να απαντήσω στο ερώτημά σας, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αναφέρει ότι 5,4 δις είναι οι επιπρόσθετες απαιτήσεις χρηματοδότησης για τη φάση μετά το 2020. Άρα τα 6,6 είναι τα χρήματα που χρειάζεται μέχρι το 2020. Δεν θα αλλάξει αυτό και δεν θα υπερπηδηθεί. Δεν θα πάμε πιο πέρα η Επιτροπή δεν θα έρθει στην αρχή την υπεύθυνη για τον προπολογισμό και θα ζητήσει, για να ζητήσει επιπρόσθετα κονδύλια μέχρι το 2020 ή για το 2020. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Το άκουσα ότι το Είτε το project αυτό έχει υποφέρει από διάφορες καθυστερήσεις και αυτό είναι ορθό. Γνωρίζουν όμως τα μέλη της Επιτροπής σας ότι τα τελευταία χρόνια η επιτάχυνση ήταν εξαιρετικά σημαντική ε, στον τρόπο λειτουργίας. Και νομίζω ότι ε, ένα στοιχείο αρκεί να αναφέρω. Πέρσι στον προϋπολογισμό πληρωμών είχαμε αύξηση κατά 268 εκατομμύρια από τα οποία δόθηκαν από την αρχή υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό τον Ιούλιο και αξιοποιήθηκαν πλήρως το έπακρο από την κοινή αυτή επιχείρηση. Βλέπετε λοιπόν πόσο έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες και τα πράγματα γενικότερα. Δεν μπορώ να προδικάσω τη μελλοντική έκβαση, μπορώ όμως να σας πω ότι... Ε, επιπρόσθετα ποσά θα αξιοποιηθούν και φέτος και θα ε, τηρήσουμε το ρυθμό με αυτή την επιταχυμένη, επιταχυμένη κατασκευή. Χάρη λοιπόν σε αυτό το θετικό κλίμα, περιμένουμε την πλήρη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο την ε, ε, απαλλαγή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να σα ρωτήσω τότε και το εξή Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο είναι τα 5,4 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτά συν τα 6 μας κάνουν 11 δισεκατομμύρια. 11 δισεκατομμύρια μέχρι πότε. Δηλαδή τα 5,4 είναι μέχρι την ολοκλήρωση, η παραγωγή πλάσματος ή μέχρι πότε για ε, να απαντήσετε παρακαλώ. Thank you. Maybe... Σας ευχαριστώ. Ίσως ε, δεν ήμουν σαφής. Είναι σαφές ότι η φάση της κατασκευής του ίτερ θα πάει πέρα από την δεκαετία του 2020, οπότε αυτό το οποίο είχε αρχικά συμφωνηθεί ως πλαφόν για την κατασκευή το 2010 προφανώς ε, δεν επαρκεί για την κατασκευή. Η κατασκευή θα συνεχιστεί πέρα από το έτος 2020 οπότε τα επιπρόσθετα λεφτά τα οποία ζητάει η Κομισιόν στην ανακοίνωση θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της φάσης ε, κατασκευής του Ίτερ που θα ολοκληρωθεί με την αρχή των επιχειρήσεων πλάσματος το 2025 σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα το οποίο ακόμα πρέπει να εγκριθεί πλήρως από την Ευρατόμ. Ελπίζω τώρα να ήμουν σαφής. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα το κατάλαβα καλύτερα. Ας ε, το δούμε λοιπόν. 2025 έχουμε το πλάσμα και μετά τι ακολουθεί. Μπορείτε να μας πείτε τι θα γίνει μετά με το ίτερ. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Αυτό το οποίο θα συμβεί μετά είναι ότι το μηχάνημα σταδιακά θα περάσει μια φάση πλήρους απόδοσης η φάση αυτή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει με την λεγόμενη λειτουργία σύνδεξης ε, το έτος 2035. Ε, Από το 2025 μέχρι το 2035 το μηχάνημα θα αποκτήσει όλον τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να αποδώσει πλήρως. Και εάν δείτε την ανακοίνωσή μας ε, πέρσι του Ιουνίου, θα δείτε ότι το κόστος ε, μέχρι το 2035 έχει καταγραφεί πλήρως. Όπως το ξέρουμε σήμερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. «5,4 δισεκατομμύρια λοιπόν μέχρι το 2035 και είναι συνολικό το πακέτο. Ε, μπορείτε να μας πείτε και νούμερα εδώ πέρα, δεν απαγορεύεται, ξέρετε. Αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Κομισιόν, ε, χρειάζομαι και άλλους πινάκες για να είμαι ακριβής με τα νούμερα, τους οποίους δυστυχώς δεν έχω μαζί μου. Έχουμε βάλει στην ανακοίνωσή μας... Α, ευχαριστώ. Τώρα μπορώ να σας πω λοιπόν αριθμούς η Κομισιόν έχει υποβάλει το πλήρες κόστος μέχρι το 2025. Πρώτα για την φάση του πλάσματος έχουμε σε τιμές 2008 είναι τιμές αναφοράς τις οποίες έχουμε προϋπολογίσει 6,6 δις έχουμε βάλει 3,9 μέχρι το 2025 αυτό σημαίνει οριστικοποίηση και ολοκλήρωση της κατασκευής. Ε, καθώς φαίνεται ότι η πρόταση για το επόμενο πι θα πάει μέχρι το 2027, περιλαμβάνεται ένα άλλο νούμερο, άλλο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος ε, του πι Για την περίοδο 2028-2035 υπάρχουν άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της κατασκευής και την λειτουργία της μηχανής. Λοιπόν, αν θέλετε το σύνολο 2020-2035 έχουμε 7,1 ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2008 που ανταποκρίνονται στα 6,6 δηλαδή ε, που έχουμε πει μέχρι το τέλος αυτής της ε, δημοσιονομικής περίοδου. Ελπίζω να ε, ήταν σαφές τώρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα Προτείνουμε λοιπόν να μας ε, φέρτε τα επικαιροποιημένα νούμερα. Ο επόμενος στον κατάλογο των ομιλητών ε, είναι ο κύριος ε, Βασίλευ για, την, για το ΣΕΖΑΡ. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον συγητή για την πολύ θετική έκθεση. Το μόνο μου σχόλιο αυτή τη στιγμή αφορά τις παροχές σε είδος που αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην παραγραφό 13 της έκθεσης. Η έκθεση μιλάει για συνεισφορές ε, σε είδος 720 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένονται από την βιομηχανία. Τα 720 εκατομμύρια είναι η συνολική αξία των έργων με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 500 εκατομμύρια με ποσοστό χρηματοδότησης 70% οπότε έχουμε 220 εκατομμύρια συνεισφορές σε είδος από τα μέλη και το 720 είναι το σύνολο αν προσθέσουμε δηλαδή τα 500 εκατομμύρια από το Eurocontrol τα συνολικές συνεισφορές σε είδος θα είναι 720 αντί για 1,2 δισεκατομμύρια. Το 1,2 περιλαμβάνει και τις ε, συνεισφορές της Κομισιόν. Αυτό γιατί χρειάζονταν να γίνει αυτή η διευκρίνηση. Για το χρονοδιάγραμμα βεβαίως μετά από τις ε, κατευθύνσεις ε, που δόθηκαν και στα μέλη το 2017. Αναμένουμε τις επόμενους μήνες να υποβληθούν τα πρώτα πιστοποιητικά κόστους, θα εγκριθούν από το Συμβούλιο και ελπίζουμε το 2017-2018 να έχουμε τις εγκρίσεις για τις ε, εισφορές σε είδος. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις είμαι στην διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ, Ιμπάνες, για στην Excel παρακαλώ. Excel. Thank you, Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την θετική αξιολόγηση. Η Excel ε, ανέλαβε δύο έργα, το ENIAC και το Artemis, ε, το 2014 και τα διαχειρίζεται και το 2015 και 16 και 17 είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια διασφάλιση για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος και η διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν να έχουμε δηλώσεις των εθνικών αρχών για το επίπεδο διασφάλισης οπότε επιτυγχάνουμε ένα υψηλότερο ποσοστό κάλυψης της χρηματοδότησης είμαστε πάνω από το 90% και θα συνεχίσουμε την διαδικασία όσο εξελίσσεται ακόμα η κληρονομιά του προγράμματος πλαισίου 7 αλλά θεωρούμε ότι τα επόμενα έτη η χρηματοδότηση η κανονική του Excel θα αντιμετωπίσει το θέμα πιο μόνιμα γιατί είναι σημαντικό αυτό για μας γιατί το Excel είναι ε, μοναδικό στο ότι έχει ακριβώς αυτή την τριμερή χρηματοδότηση και εθνική χρηματοδότηση και θα πρέπει ακριβώς να έχουμε μια κρίσιμη μάζα χρηματοδότησης ε, για να υπάρχει ακριβώς μια καινοτομία στον τομέα των ηλεκτρονικών ε, της Ευρώπης και θα στήριξουμε οπωσδήποτε και στο μέλλον και τυχόν παρατηρήσεις που θα λάβουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε τώρα στο... Στην κυρία Νόστρη, παρακαλώ. Γενική Διεύθυνση Έρευνας. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλώς ορίζουμε την έκθεση. Για βγαίνει. Συμφωνούμε. Κάποιες βελτιώσεις χρειάζονται όπως διαπιστώνετε. Κάποιες παρατηρήσεις έχω εγώ να κάνω σε σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών μέσα στην συνεργασία με το γραφείο της IMI. Ξέρετε ότι κάποια προβλήματα προκύπτουν σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα των λοιμόξεων, αλλά θα συζητήσουμε με το σχετικό γραφείο. Επίσης, τα εργαλεία πληροφορικής πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλή δυνατότητα να καλύψουμε τις καθυστερήσεις. Συνεισφορές σε είδος Αυτέ καταγράφονται από τη βιομηχανία μόνο άπαξ ετησίως και δι' το Μάρτιο. Εδώ έτσι εξηγείται η καθυστέρηση στις σχετικέ αναφορές, αλλά μέσα στον χρόνο θα συμπληρωθεί. Τελευταίο σχόλιο για ένα σχόλιο που δείχνει χαμηλό επίπεδο πιστώσεων σε σχέση με το γενικό προϋπολογισμό της ΕΜΑΗ. Εδώ αυτό οφείλεται στη γενική καθυστέρηση, στην εκτέλεση. Δηλαδή έχουμε μια φυσιολογική θα λέγαμε εξήγηση στην καθυστέρηση. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ο εισηγητής για να ολοκληρώσουμε, Brian. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και αν μου επιτρέπετε κάποιες παρατηρήσεις των συναδέλφων να τις σχολιάσω. Μίλησε στον Αστή για τη σημασία των, ε, της γλώσσας. Βεβαίως και έχει μεγάλη σημασία για να αποστείλουμε σαφή μηνύματα ε, όταν τα πράγματα πάνε καλά ή πάνε στραβά. Και πότε δεν πρέπει να ε, απολογούμαστε ή να κατηγορούμαστε για τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Για τις ερωτήσεις του κυρίου Πώς και άλλων, για το ΙΤΕΡ συγκεκριμένα, για να είναι απόλυτα σαφή τα πράγματα, έχουμε δει σημαντικέ καθυστερήσει ε, για το έργο αυτό σε ιστορική βάση. Σε ένα βαθμό απολύτω κατανοητέ καθυστερήσει, αφού εδώ χτίζεται ένα τελείω καινούριο έργο που δεν είχε προβλεφθεί στις διαστάσεις του αρχικά. Τώρα έχουμε νέα χρονοδιαγράμματα και στοιχεία για να είναι απολύτως λειτουργικό, αλλά ταυτόχρονα θα ακολουθήσει και μια φάση αφοπλισμού και πάυσης λειτουργίας. Και όσο υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία λειτουργίας, ναι, μπορεί κανείς να σταθεί, να τα κοιτάξει, να τα μελετήσει, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί και κανείς να πει ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα ποσά. Τα 5,2 όπως είπα και νωρίτερα, τα 5,2 δις είναι τα πόσα αυτά χρειαστούμε το 2020. Αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή που είμαστε δεν μπορεί κανείς να προβλέψει συνολικά ποιος θα είναι ο τελικός προπολογισμό που θα χρειαστεί, τα τελικά ποσά που θα χρειαστούν. Και αυτό προσπαθώ και εγώ να καταγράψω στην έκθεσή μου. Με σχόλια βέβαια. Παρότι αναγνωρίζω ότι υπάρχει αυτό το ποσό το οποίο ιστορικά ε, μας συνοδεύει. Έχουμε μια σημαντική όμως υπέρβαση, κατανοητή, γιατί όπως είπα ήταν τελείως καινούριο το σχέδιο, αλλά και η σημασία του δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Για τον ε, κύριο Πόχα, και τα σχόλια για το Ηνωμένο Βασίλειο και το Brexit. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει ποια θα είναι η συμβουλή του Ηνωμένου Βασιλείου ε, σε σχέση με την Ευρατόμ. Εγώ φαντάζομαι ότι θα θέλουν να συνεχίσουν και αντίστοιχα και να συμβάλλουν. Φαντάζομαι, αλλά βεβαιότητα δεν έχω. Και γι' αυτό πρέπει όλο αυτό το μεγάλο ερωτηματικό που αφορά την μοίρα της Ευρατόμ στο μέλλον με η Άνευ Ηνωμένου Βασιλείου να το συζητήσουμε, γιατί πρόκειται για ένα ακόμα, άλλη μια διάσταση κινδύνου που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Στι περαιτέρω εκθέσει. συμφωνώ με τον κύριο Πόχα σε σχέση με τη ε, σχόλια για την καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική. Γι' αυτό και αναφέρω στις εκθέσεις ότι κάθε από αυτές τι κοινέ επιχειρήσει έχει ευθύνη συνεργαζόμενη με τι άλλε να εξηγεί στο κοινό τι κάνει. Γιατί πρέπει ο πολίτης και φορολογούμενος Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζει τι γίνεται, σε ποιο επίπεδο συμμετέχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κοινέ αυτές επιχειρήσεις, οι κοινοπραξίες, πόσες θέσεις εργασίας ε, παράγονται. Άλλωστε, εάν μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με την κοινωνία, με τους πολίτες, θα έχουμε τα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα τα οποία υπογραμμίζεται. Με το ΣΕΣΑΡ έχουμε τις ε, αποτιμήσεις των εισφορών σε είδος. Θα τις δούμε. Ευχαριστώ για τα σχόλια σε σχέση με το, σφάλμα στον υπολογισμό. Και επίσης το γεγονός ότι καταγράφονται σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα οι εισφορές ανά Όλα αυτά μπορούμε να τα αντικατοπτρίσουμε. Η έκθεση όπως έχει ε, αφήνει περιθώριο σε δύο εβδομάδες συναδέλφους για υποβολή τροπολογιών με στόχο τη βελτίωση του κειμένου. Θα συνεργαστώ εννοείται με τους συναδέλφους σε αυτό το στόχο. Αλλά το κύριο μήνυμα αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, χορηγούμε την απαλλαγή, έτσι λέω εγώ τουλάχιστον, με σαφή όμως ε, ορόσημα, με σαφείς υποδείξεις που θα πρέπει στο μέλλον να τηρηθούν για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και δεν έχω μια αμφιβολία ότι θα έρθουν καλά αποτελέσματα, καλύτερα αποτελέσματα, γιατί είδαμε και με τις βελτιώσεις που καταγράφει άλλωστε και το ηλεκτρικό συνέδριο για την αντιμετώπιση των μοναπατών και τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου. Πρέπει να είμαστε όλο και πιο απαιτητικοί νομίζω. Πρέπει να είμαστε όλο και πιο απαιτητικοί και σε αυτήν την περίπτωση και νομίζω με την έκθεση αυτή στέλνουμε μια ε, καλή βάση για να χτίσουμε το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώσαμε και αυτό το θέμα τη ημερησία διάταξη και τη σημερινή συνεδρίαση. Αύριο το πρωί στι 9. Με τον Επίτροπο Όιτιγκερ. Παρόντα. Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Και καλό βράδυ σε όλους. Χαίρετε.